Cari colleghi, se per favore prendete Να καθίσετε συνάδελφοι. Ξεκινάμε σχεδόν στην ώρα μας, σχεδόν. Παρακαλώ λοιπόν να καθίσετε. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και νομίζω ότι και τα θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα απαιτούν την προσοχή μας όλων. και να εκμεταλλευτούμε και την παρουσία της υπηρεσίας διευμηνίας. Σε πάση περιπτώσει ξεκινάμε τη συνάντηση αυτή την, ε, των ε, διαφορετικών επιτροπών, τη διακοινοβουλευτική αν θέλετε συνάντηση. Υπάρχει ένας υψηλός αριθμός συναδέλφων γενικότερα. Η συζήτηση έρχεται σε καλή στιγμή θα έλεγα, είναι πολύ επίκαιρη. Διεξάγεται κατά τη διάρκεια της φάσης, στα πλαίσια της οποίας κάθε εθνική αντιπροσωπεία ουσιαστικά προσπαθεί να παρουσιάσει τις βασικές της θέσεις για τη διαπραγμάτευση. Όπως γνωρίζετε όλοι, το νομοθετικό πακέτο το οποίο θα συνοδεύει την εξωτερική υπηρεσία δεν είναι πλήρες. Ελείπει η επίσημη πρόταση για την τροποποίηση του καθεστώτος των υπαλλήλων, η οποία θα ανακοινωθεί μετά το κλείσιμο των διαπραγματεύσεων με την Επιτροπή Προσωπικού, όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Οι επίσημες επαφές όμως έχουν ήδη ξεκινήσει και έτσι και στο περιεχόμενο και για το περιεχόμενο και για τις λεπτομέρειες αυτών των επαφών θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας και τις εμπειρίες σας. Δεν θα περάσω εγώ στην ουσία της υπόθεσης, θα δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες τους οποίους έχουμε προσκαλέσει. Να μου επιτρέψετε όμως να σας μεταφέρω ορισμένε σκέψεις. Η εξωτερική πολιτική είναι ένα θα έλεγα από τα πιο σημαντικά, από τους πιο σημαντικούς τομείς ε, τους οποίους τα κράτη-μέλη επιθυμούν πάντα να ελέγχουν. Και όταν λαμβάνονται αποφάσεις στο Συμβούλιο γύρω από το θέμα αυτό, η συνένεση είναι αυτό το οποίο επιδιώκεται. Η επιλογή των θέσεων στην εξωτερική πολιτική, η επιλογή των φίλων και των εχθρών αν θέλετε, είναι κάτι το οποίο ε, εμπίπτει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Γνωρίζουμε όμως ότι οι προκλήσεις τις οποίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε καθημερινή βάση μερικές φορές ξεπερνούν, θα έλεγα, τους πόρους τους οποίους έχει στη διάθεσή του κάθε μεμονωμένο κράτος μέλος. Έτσι λοιπόν ε, θα έλεγα προκαλείται η ανάγκη συντονισμού των πολιτικών των κρατών μελών. Εφόσον δράσουμε από κοινού και με συντονισμένο τρόπο, θα μπορέσουμε να προκαλέσουμε και να επιφέρουμε καλύτερα αλλαγές οι οποίες θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά μας στον τομέα αυτό. Σαν παράδειγμα, ο ρόλος τον οποίο έχουμε αναλάβει ε, ε, στα Βαλκάνια απέναντι σε υποψήφιες χώρες όπως ε, η Κροατία. Αυτό είναι κάτι όμως που δεν εκφράζεται μόνο στη γειτονική μας περιοχή αλλά και στις πολυμερείς πολιτικές δραστηριότητές μας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συναδέλφων στα Ηνωμένα Έθνη τον προηγούμενο Νοέμβριο, ήρθε σε επιφάνεια η επιθυμία των μονίμων εκπροσώπων των κρατών μελών να αυξήσουν την δυνατότητα την οποία έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δρά αποτελεσματικά στα Ηνωμένα Έθνη και στα όργανά του. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε και τι μικτές αρμοδιότητες μπορούμε να ξεχωρίσουμε στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολούνται με τα θέματα αυτά και τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Συμβουλίου και υπολογίζοντας πάντα και κυρίως τις δυνατότητες των εθνικών διπλωματικών υπηρεσιών. Νομίζω ότι αυτή την τακτική θα πρέπει να συνεχίσουμε να την ασκούμε, να την ακολουθούμε και έτσι θα πετύχουμε μια πραγματική κεπά μια πολιτική την οποία πάντα έχουμε υποστηρίξει οι περισσότεροι από εμά. Θα πρέπει όμως σαν βουλευτές να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε αν θέλετε την διαφάνεια α, <clears throat> της υπηρεσίας αυτής. Οι αρμοδιότητες αυτής της νέας υπηρεσίας προέρχονται από τις παλαιότερες αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κάποιες επίσης διακυβερνητικές αρμοδιότητες ε, του Συμβουλίου, γιατί υπάρχουν και άλλες οι οποίες είναι αυστηρά διακυβερνητικές. Θα πρέπει λοιπόν η υπηρεσία αυτή να είναι υπόλογη και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διευρύνει τα πεδία αρμοδιότητάς του και να έρθει σε μια μόνιμη επαφή και διάλογο με την ύπατη εκπρόσωπο. Ε, νομίζω ότι πρόκειται για μια ουσιαστική κοινοβουλευτική κατάκτηση η οποία δεν είναι προς όφελος μόνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά αποτελεί θα έλεγα μια σημαντική βάση και για την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου στα πλαίσια της ΚΕΠΑ και από πλευράς των κοινοβουλίων των κρατών μελών και από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ένα πολύ σημαντικό θέμα στο οποίο αναφέρθηκαν πρόσφατα οι πρόεδροι των κοινοβουλίων στην Στοκχόλμη και θα τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά με τη Βελγική Προεδρία τους επόμενους μήνες. Εν πάση περιπτώσει έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη ευκαιρία. Μια ευκαιρία όχι μόνο να δημιουργήσουμε μια ουσιαστική πολιτική εξωτερική στην Ευρώπη, αλλά μια διαφανή πολιτική, μια πιο δημοκρατική πολιτική, μια πολιτική που να είναι πολύ κοντά στις ανησυχίες των συμπολιτών μας. Να που επιτρέψετε να σας δώσω και λίγες πρακτικές πληροφορίες τώρα για τον τρόπο με τον οποίο θα οργανωθεί η συζήτησή μας. Οι μέθοδοι που θα ακολουθήσουμε είναι αυτές τις οποίες συνήθως ακολουθούμε. Μπροστά σας έχετε όλοι φακέλους, έχετε κάποια χαρτιά μάλλον, χαρτάκια. Μπορείτε να γράψετε το όνομά σας και το κοινοβουλευτικό σώμα στο οποίο ανήκετε, όπως επίσης να σημειώσετε και το θέμα πάνω στο οποίο ε, θέλετε να πάρετε το λόγο. Ε, για να υπάρξει μια αντιπροσωπευτική συζήτηση όλων των παρόντων εδώ σήμερα θα ήθελα να σας παρακαλέσω να περιορίσετε ε, την παρέμβασή σας στα τρία λεπτά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τις εργασίες μας. με την παρέμβαση ε, του εκπροσώπου της Βαρόνης Άστον, τον κύριο Κρίστενσεν, ο οποίος θα παρουσιάσει την πρόταση για την δημιουργία της εξωτερικής υπηρεσίας. Μετά θα ακούσουμε τους κυρίους κυρίους Φερχόστατ και Μπρόκ, τους εισηγητές, και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση. Πρώτος έχει το λόγο ο κύριος Κρίστενσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να πω δύο λόγια για την σύσταση της, Ευρωπαϊκή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας πως η κυρία Καθιάστον στον λυπάται που δεν μπορεί να παραστεί αλλά δυστυχώς έχει άλλη μία επίσκεψη σε ξένη χώρα, οπότε δεν είναι σήμερα στις Βρυξέλλες. Σωστά λέτε κύριε Πρόεδρε πως είμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία αυτή τη στιγμή. Οι προσδοκίες και εντός και στους κυριότερους εταίρους μας ανά τον κόσμο για να ξεκινήσει τη λειτουργία της η υπηρεσία είναι πάρα πολύ σαφής και πολλοί από τους εταίρους μας ίσως έχουν υπερβολικές ε, προσδοκίες για το πόσο γρήγορα μπορούμε να κινηθούμε και κάθε μέρα σχεδόν μας ρωτάνε πότε θα είναι έτοιμη υπηρεσία. Νομίζω λοιπόν πως ήταν κάπως υπερβολικές οι απαιτήσεις γιατί είναι δύσκολο αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια υπηρεσία η οποία θα εξυπηρετεί την... και θα υπηρετεί την υπατή εκπρόσωπο στα τέσσερα καθήκοντα που της έδωσε η συνθήκη της Λισαβόνας όχι δύο όπως λέμε συχνά. Πέρα από αυτά τα οποία έχει ο κ. Σολάνος στο παρελθόν, δηλαδή τις πτυχές ε, εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας ε, μαζί με αυτά τα οποία είχε ως αρμοδιότητα ο Επίτροπος Εξωτερικών στο παρελθόν έχει δύο ακόμα καθήκοντα κυριάστων. Πρώτον είναι ο μόνιμος πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που από μόνο το αυτό είναι δουλειά πλήρους ωραρίου γιατί αυτό δεν σημαίνει πως ε, πρέπει μόνο να είναι παρούσα όταν ε, συνέρχεται το Συμβούλιο αλλά σημαίνει και άλλες ευθύνες ε, έναντι του Κοινοβουλίου και των κρατών μελών και κάτι ακόμα που δεν υπήρχε πριν, να δίνει μια συνοχή στην εξωτερική πολιτική, από την οικονομική, κοινωνική, την κλιματική μέχρι την πιο κλασικά νομιμή εξωτερική πολιτική. Και όλα αυτά πρέπει να τα κάνει και η υπηρεσία της. Πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου πως δεν είναι ένα παραδοσιακό Υπουργείο Εξωτερικών αυτό. Γιατί, γιατί τα καθήκοντα της ε, είπα της εκπροσώπου είναι πολύ ευρύτερα από αυτό το οποίο κανονικά ε, κάνει ένας υπουργό εξωτερικών. Έχουμε από τις πιο κλασικές πτυχές τη εξωτερικής πολιτικής μέχρι ένα οικονομικό χαρτοφυλάκιο μέχρι πράγματα όπως ε, η ηγεσία στρατιωτικών ε, ή πολιτικών επιχειρήσεων, πράγματα τα οποία δεν κάνει ένα εθνικό Υπουργείο Εξωτερικών, οπότε πρέπει να δημιουργηθεί μια δομή που θα καλύπτει και αυτά. Και τέλος, η τελευταία πρόκληση είναι να βρούμε μια δομή η οποία θα ενταχθεί στο θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει στην Ένωση. Είναι σαφές πως για πολλά από τα μέσα τα οποία χρειαζόμαστε στην εξωτερική μας πολιτική, ε, τα μέσα αυτά είναι κοινοτικά μέσα, είτε μιλάμε για την οικονομική στήριξη, ε, όπως σας είπα το κλίμα, η μετανάστευση, ε, τα πολέμησή της τρομοκρατίας, πολλά από αυτά τα πράγματα είναι στο επίκεντρο και πολλές από αυτές τις πολιτικές είναι κλασικές κοινοτικές πολιτικές, κάτι το οποίο σημαίνει πως ε, η υπηρεσία αφενός ε, πρέπει να λειτουργεί ως μια κανονική υπηρεσία της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή θα κάνει πρόταση, προτάσεις που θα υιοθετηθούν από το Σώμα των Επιτρόπων. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να καλύπτει τομείς που σήμερα σαφώς είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και όπου δεν έχει υπάρξει μεταφορά αρμοδιότητας από τις συνθήκες Λισαβόνας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πως είναι διαφορετικό το να λειτουργούμε παραδείγματο χάρη, το να λειτουργούμε τον τομέα της ε, εξωτερικής εμπορικής πολιτικής, της πολιτικής εξωτερικού εμπορίου. Δηλαδή, εάν δεν ε, μπορεί να δράσει ο αρμόδιος επίτροπος εκεί, δεν δρά κανείς. Αλλά η εξωτερική πολιτική είναι κάτι διαφορετικό. Εάν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μια κοινή λύση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε δεν υπάρχει κενό, όπως υπάρχει στην εμπορική πολιτική, γιατί θα δράσουν τα κράτη-μέλη. Οπότε η εναλλακτική δεν είναι το τίποτα, αλλά ότι θα έχουμε 27 διαφορετικές εξωτερικές πολιτικές. Οπότε θα είναι μια καθημερινή πρόκληση να έχει εξωτερική πολιτική η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι κάτι που πρέπει να καλύψουμε κατά το... την σύσταση αυτής της υπηρεσίας. Για αυτούς του λόγους είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε καλές σχέσεις με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και με την Κομισιόν, οπωσδήποτε, αλλά οπωσδήποτε και με το Κοινοβούλιο. Γιατί το Κοινοβούλιο εμπλέκεται μέσω της διαδικασίας συναπόφασης π.χ. το οποίο μπλέκεται σε οτιδήποτε φορά τα κονδύλια. Οπότε χρειαζόμαστε σε πολλού τομεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό αφορά και τη σύσταση τη υπηρεσία, γιατί αν και η βασική απόφαση για την υπηρεσία αυτή απαιτεί μόνο γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωρίζουμε πως δεν θα λειτουργήσει η υπηρεσία αν δεν αλλάξει ο κανονισμός προσωπικού, ο δημοσιονομικός κανονισμός και αν δεν έχουμε ένα προπολογισμό που θα μας δώσει αυτές τις δυνατότητες. Ε, αλλιώς δεν θα έχουμε τίποτα το ουσιαστικό. Και το συμπέρασμα λοιπόν, επειδή ακριβώς έχει το δικαίωμα της απόφαση του Κοινοβούλιο, είναι πως είμαστε σε μια de facto σχέση όπου όλα αυτά τα στοιχεία είναι πακέτο και έχει συναπόφαση εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό κατά την άποψή μας δεν σημαίνει πως πρέπει να υιοθετηθούν ε, ταυτόχρονα όλα αυτά, αλλά πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν στοιχεία από όλα τα μέρη του πακέτου όταν ε, προχωρήσουμε στην επίσημη ε, υιοθέτηση. Υιοθέτησή τους. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην κατάσταση την εξή. Είπατε εκπρόσωπος έκανε μια πρόταση. Το Συμβούλιο ε, έδωσε μια θετική γνώμη Είμαστε τώρα σε εντατικές συνομιλίες με το Κοινοβούλιο. Αναφέρατε κάποιες άτυπες διαβουλεύσεις. Νομίζω ότι περνάω περισσότερο καιρό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τελευταία παρά οπουδήποτε αλλού. Η εντύπωση μου είναι πως τα πράγματα κινούνται. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα, αλλά πλησιάζουμε και κατά την άποψή μου ε, νομίζω πως υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα τις ερχόμενες μέρες ή εβδομάδες ε, να πλησιάσουμε σε ένα πλαίσιο πολιτικής συμφωνίας και εμείς ε, θα θέλαμε να ληφθούν κάποιες επίσημες αποφάσεις πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού γιατί αν και δεν θα μπορέσουμε βεβαίω να λειτουργήσουμε πλήρως θα μπορούμε να προετοιμάσουμε τα πράγματα αν έχουμε μια βασική απόφαση επιτάπητος. Όλα αυτά πολύ σημαντικά τα θεσμικά λοιπά Αλλά βεβαίως το σημαντικότερο είναι αυτή τη στιγμή αποκτηθεί η υπηρεσία να έχουμε μια εξωτερική πολιτική ανάλογη των φιλοδοξιών μας. Νομίζω πως έχουμε την δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Είμαστε σε μια περίοδο στην οποία οι διαφορές απόψεων των κρατών μέλων δεν είναι τόσο μεγάλες. Έχουμε ξεπεράσει τις μεγάλες ε, διαφορές που είχαν τα κράτη-μέλη μετά τον πόλεμο του Ιράκ Οπότε νομίζω πως είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή συγκυρία για να πραγματοποιηθεί αυτή η φιλοδοξία. Σας ευχαριστώ. Ε, e σας ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Ήταν πολύ χρήσιμη η παρέμβασή σας. Όπως είπα πριν από λίγο, θα ακούσουμε τώρα τους δύο συνεισηγητές μας, τον κύριο Μπροκ και μετά τον κύριο Φερχόφστατ από την Επιτροπή Εξωτερικών και Συνταγματικών Υποθέσεων. Αντιστοίχως, έξι λεπτά λοιπόν για να έχουμε και χρόνο συζήτησης. Ο κύριος Μπροκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μετά από τις παρατηρήσεις του κυρίου Πρέσβη να κάνω και εγώ κάποιες παρατηρήσεις. Είμαστε σε μια φάση δύσκολων διαπραγματεύσεων, αλλά νομίζω με καλή θέληση θα έχουμε μια λύση και η καθυστέρηση βεβαίως δεν οφείλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται και λόγω των δύσκολων διαπραγματεύσεων της Κομισιόν με τα συνδικάτα δεν έχουμε καταλήξει ακόμα στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και πρέπει βεβαίως να υπάρξει και η δήλωση των οικονομικών συναπιών της υπηρεσίας αυτής. Στο Συμβούλιο είπαμε πως πρέπει να είναι δημοσιονομικά ουδέτερη Δηλαδή αυτό μπορεί να γίνει με υπαλλήλους του Συμβουλίου και της Κομισιόν, αλλά όταν το 1 τρίτο θα έρθει από τις εθνικές πρωτεύουσες, ένα τμήμα, εν αν όχι το 1 τρίτο, ε, πρέπει να υπάρχει και αναλογή χρηματοδότηση. Και θα θέλαμε να ακούσουμε ε, πώς θα τα καταφέρουμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίως αυτή τη στιγμή συμμετέχει μόνο μέσω μιας διαδικασίας διαβούλευσης. Η συνθήκη της ε, Λισαβόνας λέει πως ε, το Συμβούλιο θα συστήσει μια υπηρεσία εξωτερικής δράσης μετά από πρόταση της ΥΠΑ της εκπροσώπου με σύμφωνη γνώμη της Κομισιόν και μετά από διαβούλευση με το Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ολοκλήρωσε η διαδικασία, οπότε δεν μπορεί να ληφθεί και απόφαση του Συμβουλίου. Οπότε πρέπει να συμφωνήσουμε. Αλλά πρέπει να δούμε και άλλα δύο πράγματα. Εάν οι εθνικοί υπάλληλοι έχουν εάν είναι να ενσωματωθούν με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις σε αυτή την υπηρεσία, κάτι το οποίο θεωρώ σωστό, πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης και να έχει δικαίωμα συναπόφαση στο Κοινοβούλιο. Και αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να προσπαθήσει η αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου να βρει μια λύση. Δεύτερον, εάν πάρε δεν γίνει μια sui generis υπηρεσία τη Κομισιόν αλλά ένα ξεχωριστό θεσμικό όργανο υπηρεσία, θα πρέπει να αλλάξει το άρθρο 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. Και τότε έχει δικαίωμα συναπόφαση στο Κοινοβούλιο. Γιατί εμεί θεωρούμε πω όταν έχουμε νέε αρχέ, θα πρέπει να υπάρχει μια εγγύηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας τους. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε πως τα κράτη-μέλη δεν το βλέπουν έτσι. Πως ε, αυτό το οποίο λέει η συνθήκη ως ε, sui generis ε, είναι μια τέτοια λύση. Κοιτάξτε, εγώ επειδή ήμουν και στην συντακτική συνέλευση, αν θέλαμε κάτι τέτοιο θα το γράφαμε έτσι. Οπότε, εάν δεν είναι εντός της Κομισιόν, τότε θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς εγγύησεις κυρίως δηλαδή εγγυήσει σε ζητήματα ελέγχου. Ο έλεγχος του προϋπολογισμού, ο προϋπολογισμός και το δικαίωμα απαλλαγής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πρέπει να είναι εγγυημένα όπως συμβαίνει για την Κομισιόν. Αλλιώς θα έχουμε ένα χώρο ανεξέλεγκτο εντός της Ένωσης και όταν μετά λειτουργήσει επιχειρησιακά παρά το ότι θα είναι η λειτουργία εντός της ε, Κομισιόν δεν μπορούμε να λειτουργούμε με συμφωνίες κυρίων μεταξύ Συμβουλίου και Κομισιόν πρέπει να υπάρχει έλεγχος και πρέπει επίσης να ξεκαθαρίσουμε πως οι εθνικοί διπλωμάτες σε αυτή την υπηρεσία έχουν και υπάγονται στην ίδιες υποχρεώσεις ελέγχου με τους υπόλοιπους. Έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις, οπότε αυτό θεωρώ πως πρέπει να αποτελεί αντικείμενο εγγύησης, γιατί μέχρι στιγμής υπάρχει και ένα άλλο θέμα για το οποίο δεν είμαστε ξεκάθαροι. Εάν ο διοικητικό προϋπολογισμός τη υπηρεσία αυτή θα πάει σε ένα ξεχωριστό τμήμα, κάτι το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί ακόμα και ο υπολογισμό ΣΚΕΠΑ είναι στο τμήμα 3 της ε, Κομισιόν, τι προπολογισμού, με συγχωρείτε. Οπότε από την άλλη βλέπουμε Ε, θα έχουμε μια ένταξη εντός ε, της Κομισιόν και από πλευράς του υπολογισμού και από πλευράς διοικητικής, δηλαδή η ύπατη εκπρόσωπος ε, έχει κάποια ιδιαίτερα δικαιώματα όσον αφορά τον προϋπολογισμό και τα του προσωπικού και δεν υπάγεται πλήρως στον έλεγχο του σώματος των επιτρόπων. Επίσης ε, υπάρχει το πολιτικό ζήτημα το οποίο ανέφερε ο κ. δηλαδή το ζήτημα με ποιο τρόπο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναμειχθεί απριόρι στην ε, διαδικασία λήψη αποφάσεων. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα γίνει μέσω μιας διαβούλευσης, πώς θα έρθουν τα εμπιστευτικά έγγραφα, πώς θα γίνει ο πολιτικός έλεγχος, ποιος θα, εκπροσωπεί, ποιος θα έρχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν λείπει η κυρία Άστον, το θέμα της εκπροσώψης που είναι αποφασιστική σημασίας, όπως επίσης και το πώς ένας μόνιμος γενικός γραμματέας δεν θα κάνει de facto την δουλειά και θα είναι ανεξέλεκτος. Αυτά ως γενικές ε, παρατηρήσεις, αν θέλετε να περάσω και στις λεπτομέρειες. Μιλάμε για μια υβριδική υπηρεσία εντωμεταξύ, καθώς προσπαθεί να συμβιβάσει διακυβερνητικές και κοινοτικέ αρμοδιότητες. Και πρέπει να φροντίσουμε αυτό να μην οδηγήσει de facto στο να γίνουν οι κοινοτικέ αρμοδιότητες διακυβερνητικές. Πλην τις ΚΕΠΑ όλες οι εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 17 και 21 της Συνθήκης Λισαβόνας είναι κοινοτικέ. Πρέπει λοιπόν να ε, υπάρχουν εγγυήσει ότι αυτό δεν θα ανατραπεί για να τηρηθεί και η κοινοτική μέθοδος και τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Και θα πρέπει να δούμε εδώ πέρα αν μπορεί να διαφυλάξει τα δικαιώματα αυτά η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπροκ. Για έξι λεπτά θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο τον κύριο Φερχόφστατ. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Απλώς θα ήθελα να σας μεθυμίσω το πνεύμα και τη φιλοσοφία που διαπνέει όλους εμάς. Τον εισηγητή, τον κύριο Μπρόκ και τον ομιλούντα. Θέλουμε να υπάρχει μια υπηρεσία, όσο γίνεται καλύτερα εξοπλισμένη, όσο γίνεται πιο φιλόδοξη. Και να καλύπτει όλη την ιστορική πολιτική της Ένωσης. Ανάπτυξη, συνεργασία, γειτονία και ανθρωπιστική βοήθεια. Θεωρούμε δε ότι μόνο αν καλύψουμε όλα αυτά τα στοιχεία της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης θα είμαστε εις θέση να έχουμε μια συνοχή, συνέπεια, όπως επιβάλλεται, τόσο ώστε να μπορούμε να, πούμε ότι στη διεθνή σκηνή διαδραματίζει το ρόλο που πρέπει η Ένωση και κάνοντας όλα αυτά ασπαστήκαμε αυτή τη φιλοσοφία όπως αυτή απορρέει από την ε, ε, συνέλευση τη στεγματική του 2002 και ο κύριος Μπροκ τότε αυτό είχε βρει ως λύση για να καλύψουν την έλλειψη συνοχής και συνέπειες στην εξωτερική πολιτική. Το 2002 επομένω, αυτό ε, προέγυψε να υπάρχει ένα νέο όργανο το οποίο να μπορεί να καλύψει με αποτελεσματικότητα αυτά τα οποία απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρχει μια πραγματική, αυθεντική κοινή εξωτερική πολιτική. Και Γι' αυτό είπαμε το 2002 να έχουμε μια τέτοια υπηρεσία που να καλύπτει όλα αυτά τα οποία ε, αφορούν το Συμβούλιο, ε, δηλαδή τα διακρατικά αλλά και τα κοινοτικά όπως τη γειτονία και την ανάπτυξη. Βεβαίως η συνταγματική συνέλευση ήταν πάρα πολύ φιλόδοξη και σε εμά τώρα απόκειται να υλοποιήσουμε αυτή την ε, ιδέα. Οπότε πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι δεν αλλάζουν σε τίποτα οι αρμοδιότητες των ε, θεσμικών οργάνων, του Κομισιόν και Συμβουλίου. Ε, υπενθυμίζουμε ότι δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες αυτή η υπηρεσία που συγκροτείται. Απλώς ε, προτείνει. Στο μέλλον θα διατυπώνονται προς την Κομισιόν οι προτάσεις και προ το Συμβούλιο επίση όσον αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική. Η υπηρεσία του αυτή καθιευτεί, βεβαίω, θα πρέπει να έχει αυτονομία και και προκύπτει σαφώ ότι θα πρέπει να βρει τη θέση της ε, αυτό το όργανο στην, ε, στο, στο, στο γαλαξία των οργάνων και μια ισορροπία. Οπότε όλα αυτά τα οποία λέμε τώρα θα πρέπει να δούμε μέχρι που φτάνουν. Ε, δεν εξομοιώνεται με θεσμικό όργανο, δεν έχει τέτοιε αρμοδιότητε, δεν μπορεί να εξομοιωθεί με, τις, ε, με τα άλλα όργανα τα οποία υπηρετεί και εξυπηρετεί. Αυτή η καινούργια υπηρεσία θα διαχειρίζεται ε, στο μέλλον κάποιους κοινωτικούς πόρους, δύναμη των συνθήκων. Προβλέπεται ότι τους πόρους του χειρίζεται μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επομένως ε, προσοχή δημιουργείται εδώ κάποιο πάρα πολύ σοβαρό προηγούμενο γιατί έτσι επιτρέπεται σε μια εξωτερική υπηρεσία η οποία τώρα για πρώτη φορά εμπλέκεται στα της ε, διάθεσης εκτέλεσης του κοινοτικού προϋπολογισμού. Επομένως, αυτό που προτείνουμε είναι να υπάρξει μια θέση ε, στον προπολογισμό για αυτή την ε, υπηρεσία στο τμήμα υπαριθμών 3 που αφορά τις ε, δαπάνες, τις διοικητικές αλλά και τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες της Ένωσης. Εκεί, σε αυτό το τμήμα του προπολογισμού εντάσσονται ακόμα και όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Επομένω, σε αυτό το κεφάλαιο, στο τρίτο, εντάσσονται σχετικέ δαπάνε. Και δεν είπαμε ότι εντασσόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε αυτονομία. Ούτω ώστε να έχει αυτή η υπηρεσία το δικό τη διοικητικό προπολογισμό και, και κάνει τι ε, προσλήψεις και διορισμούς επίσης που την αφορούν. Και όσον αφορά τη διαμόρφωση τη πολιτική, είπαμε, εντάσσεται στο κοινοτικό τμήμα του θεσμικού στερεώματο. Επομένω, η μεγάλη υπηρεσία, φιλόδοξη, ούτω ώστε είπαμε ότι θα πρέπει να είμαστε ει θέση να καλύψουμε την πολιτική ανάπτυξη γειτονία και ανθρωπιστική βοήθεια. που δεν έχουν καλυφθεί ε, με άλλο τρόπο. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να έχουμε θετική κοινή εξωτερική πολιτική χωρίς να υπάρχει σύμφωνη γνώμη από τα κράτη-μέλη. Και η διαδικασία λήψη αποφάσεων ε, προβλέπει ομοφωνία. Όμως δεν μπορεί να υπάρχει κοινή πολιτική χωρίς κοινοτική προσέγγιση, χωρίς δηλαδή μια υπηρεσία η οποία μπορεί να βοηθά τον προβληματισμό ούτω ώστε να περιχαρακώνονται, να καθορίζονται τα συμφέροντα της ε, Ένωση, Δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε τις εθνικέ εξωτερικέ πολιτικές. Θέλουμε να συμπληρώσουμε το έργο τους, να το ενισχύσουμε και από αυτού είναι ξεκάθαρη η συνθήκη. Όπως ξέρετε, γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές Συμβουλίου, ε, Επιτροπής Κοινοβουλίου με την κυρία Άστον. και προσπαθούμε να δούμε πώς θα συγκροτηθεί αυτή η υπηρεσία το γρηγορότερο δυνατόν. Και ο με από τις διαπραγματεύσεις το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει όσο γίνεται. Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν τώρα τους δύο συνεισηγητές για δύο συγκεκριμένες ε, και πλήρεις ε, παρουσιάσεις. Πριν ξεκινήσει η συζήτηση θα ήθελα να ενημερώσω τους παρόντες ότι Υπάρχει μια σημαντική αντιπροσωπή από τη Σαουδική Αραβία παρούσα και εκπρόσωποι της διπλωματικής υπηρεσίας αλλά και της κυβέρνησης της χώρας. Τους καλωσορίζουμε, τους Σαουδάραβες. Υπογραμμίζουμε εδώ ότι το ενδιαφέρον το οποίο έχουν για την Ευρωπαϊκή Διπλωματική Υπηρεσία είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι ξεπερνά τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διευρύνεται και σε άλλες περιοχές, κάτι το οποίο μας ικανοποιεί. Να μου επιτρέψετε επίσης να πω ότι έχουμε εδώ ε, εκπροσώπους από 23 κοινοβούλια και 40 είναι τα μέλη από τα κοινοβούλια τα εθνικά που είναι εδώ. Έχουν ζητήσει συγγνώμη για την απουσία τους οι Ούγγροι και οι Βρετανοί βουλευτές ε, γιατί έχουν τα μετεκλογικά να αντιμετωπίσουν και επίσης δεν έχουμε εκπροσώπους Ισπανίας, Μάλτας και Αυστρίας για διάφορους λόγους. Σας καλωσορίζω όλους, θα προσπαθήσω να δώσω τη δυνατότητα να πάρουν το λόγο εναλλακτικά και στους βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα προσπαθήσω να σεβεστώ επίσης και τη γεωγραφική εκπροσώπησή τους. θα δείτε τον χρόνο τον οποίο έχετε μπροστά σας στην οθόνη σας και βλέποντας ακριβώς το πόσο χρόνος σας μένει μπορείτε να ρυθμίσετε την ομιλία σας. Θα ξεκινήσω με τον συνάδελφο Ζακ Μπλαν από τη Γαλλική Γερουσία για τρία λεπτά. Κύριε Μπλαν, έχετε το λόγο. κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη ικανοποίηση της Γαλλικής Γερουσίας να μπορέσει να συζητήσει μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την δημιουργία αυτής της εξωτερικής υπηρεσίας. Αυτή η εξωτερική υπηρεσία συνιστά θα έλεγα μια θετική και καινοτόμο ρηξικέλευθη αλλαγή θα έλεγα συνέπεια της συνθήκης της Λισαβόνας. Η Γαλλική Γερουσία έχει εκφέρει την άποψή της για τη δημιουργία αυτής της υπηρεσίας και η θέση αυτή αφορά τρεις πλευρές. Η πρώτη, Θεωρούμε ότι η εξωτερική αυτή υπηρεσία, και ακούστηκε άλλωστε αυτό προηγουμένως, θα πρέπει να είναι μια υπηρεσία sui generis, δηλαδή να απέχει εξίσου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Συμβούλιο Υπουργών, να είναι αυτόνομο στα πλαίσια της διαχείρισης του προσωπικού του και φυσικά αυτό θέτει και το θέμα του ελέγχου γενικότερα. Αυτό είναι κάτι το οποίο προέρχεται γενικότερα από την πολλαπλότητα των αποστολών της εξωτερικής υπηρεσίας. Η Γερουσία θεωρεί ότι η περίμετρος αυτής της υπηρεσίας θα πρέπει να είναι η ευρυτάτη δυνατή, να παρουσιάζει μια συγκεκριμένη συνοχή στη δράση της, και αυτό θα πρέπει να αφορά και την αναπτυξιακή βοήθεια, την πολιτική γειτονία, την ανθρωπιστική βοήθεια όπως επίσης και την ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεθνείς κρίσεις, οι οποίες δυστυχώς σοβούν. Τέλος, το ψήφισμα της Γαλλικής Γερουσίας υπογραμμίζει την μεγάλη σημασία την οποία έχει η υπηρεσία αυτή εξωτερικής δράσης και γι' αυτό θα πρέπει να έχει στενές σχέσεις με το σύνολο των κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαν και αυτό που γίνεται σήμερα όχι μόνο δηλαδή να έχει σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο χαιρετίζουμε, αλλά και με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Γιατί υπάρχει και ένα κομμάτι, αν θέλετε, της διακυβερνητικής πολιτικής και της κοινοτικής πολιτικής. Μιλάμε για ένα υβριδικό σύστημα. Αυτό επιθυμούμε και επιδιώκουμε. Αυτό, αυτή η υπηρεσία είναι, θα έλεγα, η επιβεβαίωση μιας πολιτικής βουλήσης η οποία θα κατοχυρώσει την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή. Ο ε, γερουσιαστής Μπουλό θα αναφερθεί και αυτό σε άλλες πλευρές του θέματος. Πάντως η υπηρεσία αυτή στην ουσία μεταφράζει την πολιτική βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να ξεπεράσουμε τις αντιθέσεις που υπήρχαν στο παρελθόν ανάμεσα στα κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να προχωρήσει η Ευρώπη. Ευχαριστώ ε, κύριε Γερουσιαστά. Σας συγχαίρω λοιπόν δύο φορές ε, γιατί σεβαστήκατε και το χρόνο σας. Ο εκπρόσωπος τώρα της Πολωνικής Γερουσίας για τρία λεπτά. Κέρας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας και από πλευράς της Πολωνικής Βουλής αλλά και Γερουσία, θέλω να σα ε, τονίσω τα εξή. Αυτή η πρόταση, αυτή η ιδέα του να υπάρχει μια αποτελεσματική υπηρεσία εξωτερική δράση για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πρόταση που μας ενδιαφέρει. Η Πολωνία είναι υπέρ αυτή της πρόταση και ιδέας όπως ε, έχει δημορφωθεί από τον πρόεδρο Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ε, ψηλή εκπρόσωπο που και όπω συμφωνήθηκε στις 26 ε, Απριλίου από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Και στη συνέχεια με ε, το, σχέδιο απόφαση για τη συγκρότηση αυτής τη υπηρεσία, όπου αναφέρονται πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία στα οποία συνέβαλε στη διαμορφωσή του και η Πολωνία. Πρόκειται για ένα θεσμικό όργανο που θέλουμε να συγκροτήσουμε. Έτσι θα έχουμε μια προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε και τα θεσμικά όργανα αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούν να επεκτείνουν τη δράση τους και στην σφαίρα της εξωτερικής πολιτικής. Θα πρέπει πάντως ε, να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το καινούριο όργανο ε, με τη βάση της ισότητας, της ισοτιμίας όσον αφορά όλα τα κρατημέλη και κυρίως η λειτουργία να διακρίνεται από διαφάνεια κυρίως όσον αφορά τις προσλήψεις γιατί θα πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη η γεωγραφική ισορροπία. Σήμερα προχωρούν διαπραγματεύσει και η Πολωνία χαιρετίζει ε, τις ε, δηλώσεις της υψηλής εκπροσώπου ε, σε συνεννόηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ήδη έχουν διαμορφωθεί οι αντιπροσωπείες αντιπροσωπείες των κρατών μελών υπάρχει και ο σύνδεσμος της νέας υπηρεσίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόσο ώστε να μπορεί να παρακολουθεί το Κοινοβούλιο τι γίνεται και εμείς πάντως πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ε, ασχοληθούμε περισσότερο με το πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ασκεί τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και τι θα γίνει με τον αναπληρωτή υψηλό εκπρόσωπο που ενδεχομένω θα μπορεί να αντικαθίσταται ε, από κάποιους ε, υψηλοβάθμους υπαλλήλους. Ευχαριστώ τον Πολωνό εκπρόσωπο. Από πλευράς των Ευρωβουλευτών έχει το λόγο ο κύριος Σαλαφράνκα, συντονιστής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην ΑΦΕΤ. Ε, decía el presidente de en su época de presidente de la Comisión que es muy importante en el proyecto de construcción europea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 y eh, el, la, la opinión que tiene que dar, la consulta que tiene que evacuar el Parlamento Europeo. Muchas gracias. Gracias, honorable Salafranca. Eh, pro... Ευχαριστώ κύριε Σαλαφράγκα. Ο εκπρόσωπος της Φιλανδικής Βουλής, τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Η δημιουργία, η ίδρυση θα έλεγα αυτής της εξωτερικής υπηρεσίας είναι νομίζω ένα σημαντικό βήμα το οποίο θα βελτιώσει την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν διεθνή οικονομικού εταίρου, διεθνούς οικονομικού εταίρου. Και η υπηρεσία της κυρίας Άστον και η νέα αυτή υπηρεσία νομίζω ότι έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να καταλήξουμε πάνω στα θέματα στα οποία μέχρι τώρα διαφωνούν οι διάφορες χώρες και αυτό φάνηκε και από τις ε, παρουσιάσεις που έγιναν μέχρι τώρα. Ένα τμήμα της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης δημιουργεί ορισμένα προβλήματα είναι αλήθεια, ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη. Έχουμε ζητήσει σαν παράδειγμα η υπηρεσία αυτή να είναι πλήρως υπόλογη ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι βασικές αποστολές ε, της υπηρεσίας αυτής ε, εντάσσονται στα πλαίσια της ΚΕΠΑ και εκεί οι υπεύθυνοι είναι θα έλεγα και νομιμοποιούνται δημοκρατικά να παρεμβαίνουν είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τα συμβούλια μερικές φορές κορυφής αρχηγών κρατών κτλ. Και αυτά τα συμβούλια, αυτές οι μορφές εκπροσώπησης ε, ελέγχονται δημοκρατικά από τα εθνικά τους κοινοβούλια. Λοιπόν, όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε και να μπορέσουμε να πείσουμε ε, τους ε, πολίτες ότι θα είναι ωφέλιμη η υπηρεσία αυτή, θα είναι μάλιστα και χρήσιμη για τους μεμονωμένους πολίτες ε, στα πλαίσια της λειτουργίας της ενίας ίσως προξενικής υπηρεσίας. Όλα αυτά θα βελτιώσουν την εικόνα της Ευρώπης στο εξωτερικό. Έχουμε όλοι ε, συμφέρον, κοινό συμφέρον, η υπηρεσία αυτή να μπορέσει να λειτουργήσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις. Οι συνέπειες αυτής της καθυστέρησης ε, είναι σοβαρές. Ακόμα και αν κάποιες υπηρεσίες παραμένουν διακυβερνητικές, ε, θα αλλάξουν φύση στο μέλλον στα πλαίσια αυτής της νέας υπηρεσίας. Ευχαριστώ κύριε Κόσκινο. Από τη Λετωνική Βουλή, Πάμπκης, τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε και θα ήθελα και εγώ να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Κοινοβουλίου μας και να σε ευχαριστήσω για την ευκαιρία για τη συζήτηση αυτή. Σύντομα οι σκέψεις μας τώρα για την κατάσταση, πώς βλέπουμε εμείς την εξέλιξη. Συνολικά το Κοινοβουλίο της Λετωνίας ενδιαφέρεται πάρα πολύ για να συσταθεί το συντομότερο δυνατό μια ισχυρή και ενεργή υπηρεσία εξωτερικής δράση της Ένωσης. Εμείς βεβαίως θεωρούμε πως η υπηρεσία αυτή είναι sui και θέλαμε να είναι ως το δυνατόν πιο ανεξάρτητη και στη στελέχωσή της και στον προπολογισμό της. Όσον αφορά το ερώτημά μας προς τον κύριο Κριστόφερσεν και προς την κυρία Άστον. Θα θέλαμε να ακούσουμε λίγα λόγια για το πώς σκοπεύουν να ε, στελεχώσουν αυτό το 1 τρίτο που θα έρθει από τα κράτη-μέλη και πώς θα μπορούσε αυτό να επηρεάσει τη μελλοντική εξέλιξη της υπηρεσίας Θετικά όσον αφορά δε το πεδίο δράσης, ε, συμφωνούμε με το ψήφισμα της Γαλλικής Γερουσίας και με αυτά τα οποία είπαν κάποιοι άλλοι ομιλητές που μιλάνε για συμπερίληψη ζητημάτων όπως η διεύρυνση, πολιτική γειτονία, αναπτυξιακή βοήθεια και διαχείριση κρίσεων. Νομίζω πως είναι πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και πρέπει να τις σεβαστούμε. Επίσης η Λετωνία θεωρεί σημαντικό ζήτημα μέσω της υπηρεσίας αυτής να υπάρξει μελλοντική δυνατότητα ενίσχυσης της Ευρώπης παγκοσμίω και βέβαια όταν μιλάμε για παγκόσμιο ρόλο δεν πρέπει να ξεχνάμε τους πολίτες μας και την αποξένωση μεταξύ πολιτών αφενός και Ευρωπαϊκής Ένωσης Να μην αυξηθεί αυτή η αποξένωση. Οπότε από αυτή την σκοπιά πρέπει να συνεχίσουμε να συζητάμε την δυνατότητα το προξενικό δίκτυο να ωφελήσει τους πολίτες μας, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα που πραγματικά μπορεί να βοηθήσει και σε άλλες πτυχές, όχι μόνο στην πτυχή της υπηρεσίας αυτής, αλλά και σε άλλες πτυχές της ανάπτυξης της Ένωσης. Επίσης, θα θέλαμε να τονίσουμε πως είναι σημαντικό να δούμε πιο συγκεκριμένα από την παρουσίαση του κυρίου Κριστόφερσεν πώς βλέπουν τις δυνατότητες ε, των ειδικών απεσταλμένων ε, στο πλαίσιο αυτής της υπηρεσίας. Αυτό θα ήθελα να δει το λεπτό. Ευχαριστώ. Ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη σκιώδης εισηγητής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι συνάδελφοι Μπροκ και Φερχόστατ εξήγησαν τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τις αρμοδιότητές του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως ορίζονται γύρω από το θέμα αυτό από τη συνθήκη αλλά για να πετύχει κυρίως ε, μια υπηρεσία η οποία να είναι αποτελεσματική, χρήσιμη, αλλά να σέβεται κιόλας ε, την κοινοτική μέθοδο. Εύχομαι λοιπόν να αυξηθεί το επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση στους συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων να μας θεωρήσουν φυσικούς συμμάχους γιατί θα έλεγα ότι η συνθήκη της Λισαβόνας όχι μόνο ενισχύει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά καθιστά ουσιαστικά το Συμβούλιο ένα δεύτερο νομοθετικό σώμα και έτσι του δίδει ε, πολύ πιο συγκεκριμένες ε, νομικές αρμοδιότητες σε σχέση και με τις αρμοδιότητες των Εθνικών Κοινοβουλίων. Το πρόγραμμα δράσης μας έχει ήδη, θα έλεγα, περιγραφεί όπως επίσης και οι προτάσεις ε, οι οποίες έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την οργανωτική δομή της νέας υπηρεσίας. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες ιστορικοπολιτικές που αντιμετωπίζει μια τέτοια νέα υπηρεσία. Προσπαθούμε με πραγματιστικό τρόπο να βρούμε λύσεις στις διαφορετικές απόψεις και ζητάμε να διευκρινιστούν όμως ξεκάθαρα ορισμένα θέματα τα οποία θεωρούμε πολύ σημαντικά σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εισχωρήσουμε στα πεδία αρμοδιότητας άλλων οργάνων σχετικά με την ΚΕΠΑ, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να σεβαστούμε πλήρως το άρθρο 36 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Θα πρέπει λοιπόν τα αιτήματά μας να γίνουν σεβαστά από τα άλλα θεσμικά όργανα και θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενημερώνεται σε όλες τις φάσεις επεξεργασίας και διαπραγμάτευσης των διεθνών συμφωνιών. Σχετικά τώρα με τη διαχείριση της αυτονομίας των αναπτυξιακών πολιτικών. Εμείς είμαστε υπέρ μιας φιλόδοξης, όπως είπα, εξωτερικής υπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να μπορεί να είναι σε θέση να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε επίπεδο ανθρωπιστικής βοήθειας όταν αυτό χρειάζεται. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να γίνουν σεβαστοί και οι αρμόδιοι επίτροποι και ο ξεχωριστός τους ρόλος και οι που ασχολούνται με την ανθρωπιστική βοήθεια και ε, εδώ θα ήθελα να εκφράσω την ευαρέσκειά μου για τις προσπάθειες ε, του κυρίου Κριστόφερσεν Νομίζω ότι οι προσπάθειες θα εξαρτηθεί η επιτυχία τους και από τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστεί και είπατε εκπρόσωπος για τα εξωτερικά θέματα, κάτι το οποίο θα βοηθήσει και τη λειτουργία του Συμβουλίου γενικότερα. Ευχαριστώ κύριε Γκουαλτιέρη. Ο εκπρόσωπος του Γερμανικού Bundestag για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ντάγδελεν λέγουμε, είμαι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών της Γερμανικής Βουλής. Με βάση τις διαφορετικές ε, προσεγγίσεις και συμφέροντα που κατέστησαν, νομίζω σαφή, φαίνεται πως θα πρέπει να υπάρξει ένας ρόλος της ε, Ευρώπης ε, στην διαμόρφωση της εξωτερικής αυτής ε, υπηρεσίας. Ως βουλευτής κυρίαρχου κράτους είναι και για εμένα πάρα πολύ σημαντικό η εξωτερική πολιτική να συνεχίζουμε να συναποφασίζουμε την εξωτερική πολιτική στην Γερμανική Βουλή και να μην πάει η εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρόπον την Και βέβαια αυτό σχετίζεται με την σύλληψη της ε, υπηρεσίας αυτής, καθώς εδώ πέρα πηγαίνουμε προς μια εξασθένηση της αποφάσεως ε, όπως ε, αναφέρει και η απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, μια εξασθένηση των ε, δικαιωμάτων των κοινοβουλίων, ειδικά όσον αφορά στρατιωτικές επιμάσεις. Οπότε έχουμε εδώ πέρα μια... Το έχουμε μια εξασθένηση των εθνικών πολιτικών, οπότε πρόκειται για κάτι το οποίο μας ανισχύει και είναι κάτι το μοναδικό στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας δικαίως δεν έχουν συγχωνευτεί σε ένα. Να μην πω δε για το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτός ο διαχωρισμός λοιπόν διπλωματικών και στρατιωτικών δομών αποτελεί ε, πυλώνα του δημοκρατικού μας κράτους και σε εμά και σε άλλες χώρες. Οπότε υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα, ξεκινώντας από το πώς θα υπάρχει αποτελεσματικός δημοκρατικός και κοινοβουλευτικός έλεγχος αυτής της υπηρεσίας, μέχρι το πόσο περισσότερο θα κοστίσουν αυτές οι υπηρεσίες δεδομένης δε της τεταμένης οικονομικής κατάστασης στα κράτη-μέλη και στην ίδια την Ένωση. Αυτό αναρωτιόμαστε ως βουλευτές πόσο θα κοστίσουν ε, επιπλέον όλα αυτά. Αυτό το οποίο δεν χρειάζεται η Ευρώπη είναι άλλη μια στρατιωτικοποιημένη υπηρεσία που θα κοστίζει δισεκατομμύρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Ντάγκ λέει ο Πρόεδρος και τώρα το λόγο έχει ο Ριμπέιρο Κάστρο, ε, από την Πορτογαλία. Έχει για τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κατόπιν των όσων ακούσαμε από τον κύριο Κριστόφρασεν, εγώ θα ήθελα να σας πω το εξή. Η συγκρότηση αυτής της ε, υπηρεσίας τελικά έχει πάρει περισσότερο χρόνο από όσο στην αρχή ε, προβλεπόταν. Βέβαια αυτό δεν μας προξενεί έκπληξη γιατί πρόκειται περί περίπλογης και δύσκολης υπόθεσης. Ε, οπότε καλύτερα, επομένως, ε, κανείς να σπέβδει βραδέας. Να μην βιαζόμαστε και κάνουμε τα πράγματα στο γόνατο. Από την άλλη μεριά, θα πρέπει να εξετάσουμε τι γίνεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίω και θα πρέπει να κατοχυρώσει τι αρμοδιότητέ του και να τι οριοθετήσει. Όμω, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τι σχετικέ διαβουλεύσει. Γιατί τώρα ε, βρισκόμαστε σε συναπόφαση. Αφού το προβλέπει η συνθήκη, αυτό θα πρέπει να τηρηθεί. Επομένως, οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να ενεργήσουν αντίστοιχα κατά την σχετική διαβούλευση. Τώρα έχω κάποιες ερωτήσεις για τον κύριο Κριστόφερσον. Θεωρείτε ότι η υπηρεσία της κυρίας Άστον μπορεί να προγραμματίσει και διεξαγάγει επισκέψεις στα εθνικά κοινοβούλια. Επίσης, όπως είπε η συνάδελφος από τη Γερμανία, έχουμε και εμείς κάποιο προβληματισμό όσον αφορά το δημοκρατικό έλεγχο του του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, τι θα γίνει με τον έλεγχο τον οικονομικό. Θα πρέπει επομένω η κυρία να έρθει σε επαφή με τις επιτροπές εξωτερικών υποθέσεων των Εθνικών Κοινοβουλίων και να διασκεδαστούν οι σχετικές αμφιβολίες και επιφυλάξεις. Κάτι άλλο τώρα. Πεςτε μας ακριβώς και συγκεκριμένα από ποιους θα απαρτίζεται αυτή η υπηρεσία. Είπαμε ότι το 1 τρίτο θα διορίζεται από τα κράτη-μέλη. Αυτό πώς προχώρησε, πώς, πώς βαδίζει. Τέλος. Θα ήθελα να σας πω ότι θεωρώ πως η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ορθώς καλύπτει τόσα πολλά θέματα όπως εξωτερικό εμπόριο, όπως ανθρωπιστική βοήθεια και αυτό είναι σωστό όχι μόνο γιατί αυτά είναι θέματα εξωτερικής πολιτικής αλλά γιατί θεωρώ ότι είναι σωστό μια τέτοια υπηρεσία εξωτερικής υπηρεσίας να, να, να, να, να μην έχει κολοβωμένη την αρμοδιότητά της και τη δράση της για να μπορεί να καλύψει αυτά τα θέματα ε, προσοχή το εξωτερικό εμπόριο είναι κοινοτική αρμοδιότητα και βέβαια θα πρέπει κάπως να αξιοποιηθεί η αποκτηθήσα εμπειρία από όλα αυτά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Μπέο Κάστρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ομάδα μου τους Πρασίνους. Είναι σημαντικό αυτή η κοινή εξωτερική υπηρεσία να είναι μια φιλόδοξη υπηρεσία η οποία θα εκπληρώνει τους στόχους της και σε άλλες υπήρους. Δηλαδή την καταπολέμηση της φτώχειας και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό σημαίνει του χάρη πως υποστηρίζουμε αυτό το οποίο είπαν κάποια μέλη εθνικών κοινοβουλίων, δηλαδή το ότι οι υπηρεσίες αυτές ή προξενικές θα πρέπει να εξυπηρετούν από κοινού τους πολίτες. Ήμουν 10 χρόνια βουλευτής στο Εθνικό Κοινοβούλιο της Αυστρίας και η σημερινή στη σημερινή συνεδρία θεωρώ πως είμαστε σύμμαχοι εθνικοί βουλευτές και ευρωβουλευτές στη δημιουργία αυτής της υπηρεσίας και κάποιοι φόβοι που άκουσα πως ε, τα εθνικά κοινοβούλια χάνουν επιρροή δεν ε, με βρίσκουν ε, σύμφωνοι και στη συνάδελφο από τη Γερμανική Βουλή που λέει πως δεν θα αποφασίζουν τα εθνικά κοινοβούλια για στρατικές αποστολές αυτό απλά δεν ισχύει, δεν ισχύει, όχι Α, απλά δεν ισχύει, συγγνώμη. Όχι, ε, εγώ έχω το λόγο, σας το λέω. Είμαι των πρασίνων μέλος, με ανισχύει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Εξακολουθούν τα εθνικά κοινοβούλια να αποφασίζουν τώρα για τα επί Το ότι θα υπάρχει μια υπηρεσία που θα ασχολείται με ζητήματα γειτονίας και αναπτυξίου τίποτα άλλο πρέπει να ξεκαθαρίζει και για εμάς πως ε, θα παραμένουν οι οικονομικές αρμοδιότητες ανάπτυξης στον Επίτροπο Ανάπτυξης. Τώρα κάποια σημεία που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Χρειαζόμαστε μια γενική διεύθυνση εδώ πέρα για διαχείριση κρίσεων, ε, πρόληψη συγκρούσεων και οικοδόμηση ειρήνης. Το προτείνει αυτό η συνθήκη της Λισαβόνας, οπότε θα πρέπει να είναι εντός της υπηρεσίας κατόπιν. Θα πρέπει να δούμε το πώς θα εφαρμοστεί η ισότητα ανδρών και γυναικών σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή στην επιλογή του προσωπικού. Γνωρίζουμε πως ειδικά στην εξωτερική πολιτική και στα κοινοβούλια δυστυχώς δεν έχουμε αρκετή παρουσία γυναικών, σημαίνει Δηλαδή, εντάξει, η κυρία Άστον εδώ πέρα είναι μία σύμμαχός μας, πρέπει να το ξεκαθαρίσει, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μία ξεκαθαρή, ξεκαθαρή πολιτική ενσωμάτωση των πολιτικών ισότητας. Επίσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα που το ανέφερε ένα συνάλφος από την αρμόδια επιτροπή, πράγματι χρειάζεται αυτά να εδρεωθούν ε, κεντρικά στην ε, υπηρεσία αυτή. Αναφέρεται επίσης στην, ε, στο άρθρο 21 όπως επίσης και στα βασικά σημεία των αντιπροσωπείων κατά τα λοιπά. Υποστηρίζουμε τις απαιτήσεις των κυρίων Μπροκ και Φερχόφστατ, κυρίως ε, όσον αφορά το τμήμα 3 του προϋπολογισμού, αν είναι να μιλάμε για συνοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τον λόγο ο κύριος Νταλάρας, η κυρία Ντελάρα από, το, τη Βουλή των Ελλήνων. Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περίοδο με σημαντικές γεωπολιτικές ανακατατάξεις και μέσα στη γενική κρίση, όπως είπε και η προλαλή σας συνάδελφος, μπορεί να παίξει ρόλο σε θέματα όπως την καταπολέμηση της φτώχειας. Αναφυσβήτητα αποτελεί ένα στίχημα για την Ένωση μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ωστόσο, σαν εκπρόσωπος του ελληνικού, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα ήθελα να επισημάνω ορισμένα στοιχεία. Η νέα υπηρεσία θα πρέπει να λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στη στελέχωση αλλά και στον καθορισμό των αρμοδιοτήτων. Γι' αυτό και το οργανόγραμμα θα πρέπει να καταγραφεί επακριβώς αυτή την απόφαση. Ε, ε, σε παρένθεση λέω ότι συμφωνούμε αρχικά με την πρόταση της ισόρροπης εκπροσώπησης, αν τρίτο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν τρίτο κράτη-μέλη και ένα τρίτο από το Συμβούλιο. Επιπλέον στο νέο αυτό διοικητικό σώμα θα πρέπει να υπάρξει σεβασμό στην αρχή της γεωγραφικής κατανομής σε σχέση με τη στελέχωση ώστε όλα τα κράτη-μέλη να εκπροσωπούνται αναλογικά και να μην έχουμε αποκλεισμού. Ιδιαίτερα επίση σημαντικό για την αποτελεσματική λειτουργία τη νέα υπηρεσία είναι η διαμόρφωση μηχανισμών γρήγορη και αποτελεσματική διαβούλευση μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κρατών μελών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που τελικά έχει το δημοσιονομικό έλεγχο μέσω τη διαδικασία τη συναπόφαση. Η αποφυγή τριβών, επικαλύψεων, αρμοδιοτήτων πρέπει να αποτελεί πρώτο στόχο για όλου, ώστε να μην έχουμε φαινόμενα διγλωσία συγχύσεων, καθυστερήσεων στη λήψη και υλοποίηση αποφάσεων που τελικά υπονομεύουν όχι μόνο τη λειτουργία αυτή τη νέα αξιόλογη υπηρεσίας αλλά και τη διεθνή παρουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ επίσης σκόπιμο να αναφέρω την ανάγκη συνεργασία τη νέα Υπηρεσία, όχι μόνο με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό θα αποτελέσει το ανακρογωνιαίο λίθο για την καλύτερη δυνατή λειτουργία αλλά και την ανάδειξη του ρόλου της νέας αυτής υπηρεσίας που μπορεί να παίξει, επαναλαμβάνω, ένα σημαντικότατο ε, ρόλο στα, στα διαρκώς ανακύπτοντα θέματα που έχουν σχέση με την κρίση την οποία βιώνουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Νταλάρα. Το λόγο έχει ο Λαμπέρτο Ντίνι, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Ιταλικής Γερουσίας. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Βέβαια, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε όλοι το, το, το προνόμιο και την τύχη να μπορούμε να μιλήσουμε με την μετρική μας γλώσσα. Όμως, θα σας μιλήσω στα αγγλικά, διότι είναι μία από τις δύο γλώσσες εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. θέλω να σταθώ σε αυτά τα οποία είπαν οι κύριοι Κρίστοφσεν, ε, Φερχόφστατ και Μπροκ. Και πρώτα-πρώτα σας αναφέρω ότι άπαξ και μπορέσουμε να έχουμε συγκροτημένη την εξωτερική υπηρεσία. Αυτό δεν πάει να πει ότι θα έχουμε και εξωτερική πολιτική. Ποιος θα τη διαμορφώσει. οι υπάλληλοι αυτή τη εξωτερική υπηρεσία θα τη διαμορφώνουν ή απλώ θα είναι διεκπαιρεωτικό ο ρόλο του περιπτικός για τις ε, αποφάσεις που θα λαμβάνονται αλλού, ας πούμε, ε, στο Συμβούλιο, εκεί όπου η κυρία Άστον θα αναφέρεται. Επίσης, δεύτερον, συμφωνούμε εις το ότι πρόκειται για μια υπηρεσία ιδιότυπη σου γένερης. Δεν είναι ένα νέο θεσμικό όργανο, είναι μια υπηρεσία ε, αυτεξούσια, αυτάρκης, αυτόνομη όσον αφορά προσωπικό και πρεκοδότηση προπολογισμό. Και πολύ σωστά τα είπε ο κύριο Μπροκ όσον αφορά την υποχρέωση ε, λογοδοσίας και δημοκρατικού ελέγχου. Δεν αρκεί μια συμφωνία κυρίων μεταξύ Συμβουλίου, υψηλή εκπροσώπου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει ξεκάθαρα αυτό να διατυπωθεί εις κάποιο έγγραφο. Δεν λέω ότι είναι θέμα διοργανικό, αλλά θα πρέπει όμως πάρα πολύ συγκεκριμένα να προβλέπετε. Για παράδειγμα, στην ε, διακήρυξη δήλωση της ψηφιακής εκπροσώπου όσον αφορά το δημοκρατικό έλεγχο, εντάξει, εδώ λέει ότι ε, εκείνη πρόκειται να συμβουλεύεται το κοινοβούλιο όσον αφορά βασικά σημεία κλπ. Αυτό θα πρέπει να επισημοποιηθεί σε κάποιο έγγραφο, το οποίο και θα διέπει τις σχέσεις των οργάνων μεταξύ Τώρα, συγκεκριμένα όσον αφορά αποστολές. Αναφέρεται εδώ ότι το Κοινοβούλιο πρόκειται ε, να διαβουλεύεται με την υπηρεσία όσον αφορά τις αποστολές που θα χρηματοδοτούν από τον κοινοτικό προπολογισμό. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει για όλες τις αποστολές ε, να είστε τη γνώμη του Κοινοβουλίου. Ας πούμε, οι στρατιωτικέ αποστολέ, οι οποίες πρικοδοτούνται από τα κράτη-μέλη και δεν ε, αποτελούν τμήμα ή, αποτελούν τις εξωτερικές ε, εξωτερική δράση. Επομένω, νομίζω ότι όλε οι αποστολέ θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαβούλευση με το Κοινοβούλιο. Επίσης, είπε ο κύριος Μπρόκ, σε σχέση με ε, τον πολιτικό έλεγχο, όταν δεν, όταν δεν υπάρχει κάποιος φιλός εκπρόσωπος, ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αυτός είναι ο, ο αιρετός άρχον. Αυτός θα πρέπει να έρχεται εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο και να γίνεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και η συνεννόηση με το Κοινοβούλιο. Κύριε Βερχόφστατ, επίση συμφωνούμε στο ότι αυτή η υπηρεσία θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο φιλόδοξη. Και να είναι ευέλικτη, μην είναι ένα και όχι μόνο για λόγου εξόδων δαπανών, όπω είπε η Γερμανία συνάδελφο, αλλά και για λόγου αποτελεσματικότητα. Διότι θα πρέπει ε, αυτή η υπηρεσία να δίνει καθημερινέ γραμμέ και όχι να υποκαθιστά την λειτουργία και οργάνωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, όλε οι εξωτερικέ υπηρεσίε τη Κομισιόν θα πρέπει, θα πρέπει να συνεχίσουν να υπάγονται ή στην Κομισιόν και να μην υπαχθούν στην καινούργια υπηρεσία. Χρειαζόμαστε συντονισμό. Η εκπρόσωπο τελικά είναι αντιπρόεδρο τη Κομισιόν. Επομένω, ψηλή εκπρόσωπος μπορεί να ασχεί τα καθηκοντά από την υπάρχουσα θέση τη, χωρίς να πρέπει να φτιάξουμε μια, μια, μια μεγάλη και υπηρεσία χωρίς καμία ευελιξία. Επόμενος, να δούμε τελικά ποιοι θα ε, αποσπαστούν σε αυτή την υπηρεσία. Χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε διπλωμάτες. Όπως γίνεται παντού θα χρειαζόμαστε μια διπλωματική σχολή και για του Ευρωπαίου διπλωμάτε. Ο κύριος Νταφ για τρία λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, η συνθήκη θα μας ενθαρρύνει να βελτιώσουμε την ποιότητα και την συχνότητα της ε, συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοβουλευτικών επιπέδων. Δεν είναι κανονιστική και πρέπει να ε, ερχόμαστε συχνά σε συνεννόηση πριν καταλήξουμε σε, στην κατάλληλη συνταγή, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα φόρουμ το οποίο θα είναι το κατάλληλο για να δεχόμαστε και να εξετάζουμε τον πρόεδρο Φαν Ρόμπαϊ όπως και την κάθε Άστον γιατί και οι δύο έχουν ευθύνη για την ΚΕΠΑ. Αλλά κάποιοι συνάδελφοι νομίζω ήταν επιλεκτικοί στην ερμηνεία της συνθήκης. Η κάθε άστον δεν είναι ε, η μόνη υπεύθυνη για την ΚΕΠΑ αλλά είναι υπεύθυνη και για τον συντονισμό όλων των εξωτερικών δραστηριοτήτων της Ένωσης και η υπηρεσία εξωτερικής δράσης στόχο έχει να υπηρετεί την καθιάστον. Πρέπει λοιπόν να βλέπουμε συνολικά την συνθήκη. Ο κύριος Ριμπέρο Ικάστρο Φάνηκε είπε πως ε, η κυρία Καθιάστον θα πρέπει να πάει σε 27 εθνικά κοινοβούλια. Μπορώ να του πω πως ε, αυτό δεν είναι καθόλου πρακτικό. Δηλαδή τις ζητάμε να είναι σε κάθε γωνία της Ιφιλίου και στις Βρυξέλλες και είναι αδύνατο για αυτήν να εκπληρώσει σωστά τα καθήκοντά της και ως προς την κοινοβουλευτική δημοκρατία εάν ε, είναι να τρέχει σε 27 εθνικά κοινοβούλια και στο, Εθνικό, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε θα πρέπει να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε το ποια είναι η κατάλληλη προσέγγιση για να λυθεί αυτό το ζήτημα της κοινοβουλευτικής συνεργασίας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τηλιανίδης. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση κύριε Πρόεδρε. Ίσως μετά την παρέμβαση του κυρίου Ντίνη πολύ λίγα να μπορούν να λεχθούν απλώς ως συμπληρωματικά. Όμως φαίνεται από τη συζήτηση ότι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η υπηρεσία θα είναι αυτόνομη, σου generis κατάσταση. Θα την κρίνουν τρία πράγματα η αποτελεσματικότητα, η συνοχή στη δράση και να έχει πολιτικό ρόλο. Προς Θεού, εάν παραμείνει αποκλειστικά και μόνο στην ανθρωπιστική βοήθεια, την οποία εκτιμώ βαθύτατα, νομίζω ότι δεν θα επιτελέσει το ρόλο της. Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα, οι προτάσεις και του κυρίου Προκ και του κυρίου Φέρχοσταρτ και τώρα του κυρίου Ντίνη έχουν ήδη δώσει το πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να φτάσουμε για να έχουμε αποτελεσματικότητα. Η συνοχή στη δράση έχει σχέση όντως και με τα εθνικά κοινοβούλια και με, τις, και με τα Υπουργεία Εξωτερικών των κρατών μελών. Στο δικό μας κοινοβούλιο έχει συζητήσει ήδη το θέμα διεξοδικά και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι προτάσεις όπως κατατίθενται για την ισορροπία των τριών μερών είναι μια καλή αρχή. Υπάρχει όμως περίπτωση να βρεθούμε στο δίλημα κοινοτική versus διακυβερνητική. Αυτό το δίλημα θα μπορεί να το συμπληρώνει και να το λύει η διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει και τον ρόλο εκ για το δημοκρατικό έλεγχο μέσα στην κρίση του ευρώ που περνούμε όλοι μας. Μια τέτοια υπηρεσία μπορεί να δώσει τέτοιο πολιτικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα βοηθήσει ακόμη και την εικόνα της ως οικονομική δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Στυλιανίδη από την γερουσία της Τσεχίας ο κύριος Βόντρα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι σημαντικό το να εμπλέγω σε αυτή τη διαδικασία τα εθνικά κοινοβούλια. Ήταν καλή ιδέα. Όχι δεν λέω ότι τώρα θα μπορέσει και πρέπει τώρα η υψηλή εκπρόσωπος να πάρει βάρνα τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά νομίζω τον έρχεται εδώ, είναι θετικό. Και πρέπει να σας πω ότι εν γέννη συμφωνούμε με τα όσα έχουν προταθεί. Και είναι πάρα πολύ σημαντικές παράμετροι, πρώτα-πρώτα, το τι θα γίνει σε αυτήν την ισορροπία δυνάμεων, αλλά και την κατανομή του προπολισμού των εξωτερικών οργάνων. θα πρέπει να λειτουργήσει όπως λειτουργεί κάθε δημοκρατικό όργανο στη δημοκρατία. Ξέρουμε ότι υπάρχει χρονική πίεση και θα πρέπει και εμείς να αποδείξουμε ότι έχουμε μια αυθεντική εξωτερική πολιτική και ότι είναι σημαντικός παίκτη τη εθνική Κοινή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, δεν είναι θέμα ποσότητας και ταχύτητα είναι ποιότητα. Τώρα θέλω να σας πω τα εξή. Όσον αφορά την εκπροσώπηση, καταρχήν συμφωνώ με τον Λαμπέρτο Θα πρέπει να έχουμε αγγλικά ή γαλλικά γλώσσα εργασία, τόσο ώστε να ε, υπάρχει καλύτερη συνεννόηση. Επίσης, να χωνέψουμε ότι δεν είμαστε εμείς από τη μία και απέναντι η υπηρεσία, εμείς και οι άλλοι, ότι είναι δική μας η υπηρεσία. Επίσης, έχω την αίσθηση ότι οι Γάλλοι αισθάνονται ότι αδικούνται, δεν εκπροσωπούνται επαρκώς. Όμως, για κάτι να σκεφτείτε, εμείς, τα νέα κράτη-μέλη και άλλοι, να το θέμα της γεωγραφικής ισορροπίας στην εκπροσώπηση. Μπα και είχαμε πειρασική κυβέρνηση και γι' αυτό δεν προσωπηθήκαμε πάντως. Ας ισχύσει αυτός, αυτή η παράμετρος, η μέθοδος του Κίνοκ, αυτό το οποίο έγινε τότε που έγινε η, το 2004 με την ε, διεύρυνση. Ούτως ώστε κάπως τουλάχιστον ε, υπάρχει κάπως, κάπως δίκαιη εκπροσώπηση παρά το ότι απέχουμε πάρα πολύ από εκείνο το οποίο θα θέλαμε να δούμε. Επίσης και πάλι σχέση με την ε, διεύρυνση. Εάν θέλουμε να είμαστε σοβαροί όσον την πολιτική της διεύρυνσης, θα πρέπει να θεωρήσουμε την διεύρυνση εσωτερική υπόθεση και όχι εξωτερική. Ε, mm. ε, Ευχαριστώ κύριε Βόντρα. Το λόγο έχει ο κύριος Τάνοκ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η δική μου ομάδα έχει μια σχετικά μειονοτική άποψη, μειοψηφική καλύτερα θα έλεγα άποψη. Εκπροσωπώ τους Βρετανούς συντορητικούς. είμαστε κατά τις συνθήκες της Λισαβόνας και είμαστε κατά και της εξωτερικής υπηρεσίας. Εξελισσόμεθα όμως, τώρα είμαστε σε συνασπισμική κυβέρνηση και έχουμε γίνει ξαφνικά πολυπραγματιστές. Πιστεύουμε ότι η εξωτερική υπηρεσία θα πρέπει κυρίαρχα να είναι ε, διακυβερνητική και να ελέγχεται από το Συμβούλιο, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει σχέση με την ΚΕΠΑ, που είναι ο βασικός της, θα έλεγα, συστατικός λόγος και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να την ενσωματώσουμε σε αυτήν την υπερεθνική μορφή την οποία έχει αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει βέβαια και πέρα της ΚΕΠΑ θα ασχολείται με θέματα ανάπτυξης, ανθρωπιστικής βοήθειας, διεύρυνσης και γενικά θα πατήσει σε αρμοδιότητες παλαιότερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ξέρω ότι η ανθρωπιστική βοήθεια είναι κάτι στο οποίο ε, ε, θα έλεγα επιμένει ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκεί θα εισχωρήσει η νέα αυτή εξωτερική υπηρεσία. Αλλά από την άλλη δεν δημιουργούνται μέσω της συνθήκης της Λισαβόνας νέες αρμοδιότητες στα πλαίσια της ΚΕΠΑ θα έλεγα για τα κοινοτικά όργανα, αν και υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων σε επίπεδο ας πούμε ρύθμισης οργανωτικής, σε επίπεδο πολιτικής προσωπικού κτλ. και έχει de facto πλέον αποκτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, την δυνατότητα ελέγχου σε οποιαδήποτε φάση των δραστηριοτήτων ε, της ε, εκπροσώπου μας στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Βλέπουμε λοιπόν ότι πλησιάζει σε επίπεδο αρμοδιοτήτων τις αρμοδιότητες τις οποίες έχει το Αμερικανικό Κογκρέσο όταν επιβεβαιώνει τους διορισμούς τους οποίους προτείνει ο πρόεδρος της χώρας. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαριστούν τα προβλήματα αυτά και να καθοριστεί επίσης και το θέμα του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Εμείς πιστεύουμε σαν πολιτικό κόμμα ότι θα πρέπει να μην διευρύνουμε το πεδίο δραστηριότητας της συγκεκριμένης υπηρεσίας σε τέτοιο επίπεδο έτσι ώστε ε, ε, να καλύψει όλες τις αρμοδιότητες ε, και θα πρέπει και το θέμα της γλωσσομάθειας να αντιμετωπιστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην επιλέγεται ε, συστηματικά ένας ε, διπλωμάτης από οποιαδήποτε χώρα ε, επειδή έχει πολλές γνώσεις όταν πρόκειται όμως να βοηθήσει στη σύναψη μιας συμφωνίας με την Κίνα όπου αυτό το οποίο θα μετράει θα είναι η γνώση της κινέζικης γλώσσας. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι στις απαιτήσει τις οποίες θα έχουμε. Ξέρουμε επίσης ότι αυτοί που θα λαμβάνουν αποφάσεις μερικές φορές θα είναι δύσκολο να καθοριστούν γιατί ε, και οι ε, αρμόδιοι ε, και σε επίπεδο Συμβουλίου και σε Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πάρα πολύ συχνά δεν θα είναι παρόντες για να παίρνουν τις αποφάσεις οι οποίες χρειάζονται. Θα πρέπει ιδιαίτερα μετά από τη διέλυση της διακοινοβουλευτικής συνέλευσης της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης να ενεργοποιηθούν τα εθνικά κοινοβούλια έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε την αρχιτεκτονική της κοινή εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επόμενη δεκαετία. Βάλκενς από την κάτω βουλή της Ολλανδίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μας δίνετε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε σκέψεις εδώ πέρα για την σύσταση της ευρωπαϊκής αυτής ε, υπηρεσίας. Έχουμε και εμείς κάποιες ερωτήσεις για την κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών μεταξύ της ΣΥΠΑ, της εκπροσώπου της υπηρεσίας και του Επιτρόπου Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Η Βουλή μας θεωρεί πως μια συνεκτική και ολοκληρωμένη εξωτερική πολιτική είναι ουσιαστική για την Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο, αλλά εντός ενός διακυβερνητικού πλαισίου, με σεβασμό για τις αρμοδιότητες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Είναι σημαντικό να παραμείνει η διοργανική ισορροπία. Τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να μπορούν να επηρεάζουν την κατάσταση μέσω των κυβερνήσεών τους. Σημαντικό είναι να πούμε πως στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας η Ολλανδία έχει φιλοδοξίες και θέλουμε να συνεργαστούμε με τα ευρωπαϊκά όργανα. Θέλουμε να είναι επιτυχημένη αυτή η υπηρεσία επί τη βάση της συνεργασίας με αφετηρία τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας και με το δικαίωμα συναπόφασης και του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών και των Κοινοβουλίων. Μιλάμε δηλαδή πρακτικά για την αποτελεσματική λειτουργία της ε, υπηρεσίας η οποία δεν θα πρέπει να εξαντληθεί μόνο σε έναν καυγά για το ποιος θα έχει την εξουσία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βάλκεντς. από τη Ρουμανική Βουλή ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Επιτρέψτε να μιλήσω στην μητρική μου γλώσσα. Συνεχίζει στα ρουμανικά. Από πλευράς της ε, γερουσίας τη χώρα μου θεωρούμε ότι πάρα πολύ καλή ιδέα ήταν να οργανωθεί αυτή η συνάντηση. Το Βουγουρέστη θεωρεί ότι αυτή η υπηρεσία θα πρέπει να είναι λειτουργική. Να βοηθάει, να ακούγεται με μία φωνή Ευρωπαϊκή Ένωση στην διεθνή σκηνή. Όμως θα πρέπει να διέπεται η λειτουργία αυτής της ε, υπηρεσίας από τα εξή. Θα πρέπει να διακρίνεται από αυτονομία θα πρέπει να έχει τον δικό της προϋπολογισμό. Θα πρέπει να έχει απολυστική αρμοδιότητα για το προσωπικό της. Και όλα τα κρατημέλη θα πρέπει να εξυπηρετούνται και να έχουν ε, καλή συνεργασία με αυτή την υπηρεσία. Να είναι δυνατόν να υπάρχουν ε, και διμερείς σχέσεις αυτής της υπηρεσία με τα κράτη-μέλη και γενικά η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διακρίνεται περισσότερη συνέπεια. Συμφωνούμε με το, αυτά που ακούστηκαν ότι δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τον διορισμό του προσωπικού της ε, υπηρεσίας. Θα πρέπει να ισχύσει κάποια γεωγραφική ισορροπία στην επιλογή των υπαλλήλων και να υπάρχει ισοτιμία όσον αφορά δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών των ε, υπαλλήλων. Θα πρέπει να προχωρήσουμε ταχαίως στην συγκρότηση της υπηρεσίας, να υπάρχει ένας διορθωτικός προπολογισμός που να πρεκοδοτεί στην υπηρεσία αυτή και για να δούμε τώρα τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την υπόθεση. Θα πρέπει να πετύχουμε ισορροπία μεταξύ των εθνικών από τη μια και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την άλλη. Γιατί όλοι μπορούν να συμβάλλουν στην συγκρότηση αυτής της ε, υπηρεσίας να λάβει υπόψη τι λένε οι συνθήκε. Δημοκρατική νομιμότητα βέβαια έχουν και τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τελικά το τι θα κάνουμε θα πρέπει να διέπεται από την επιθυμία μας να συγκροτηθεί μια αποτελεσματική υπηρεσία. Να λάβουμε υπόψη την πολιτική της ε, γειτονίας. Ε, βεβαίως και η διεύρυνση θα πρέπει να περνάει μέσα από την καινούργια υπηρεσία, να έχουμε στρατηγική, να έχουμε πραγματική πολιτική και όχι μόνο τεχνοκρατική αντίληψη της εξωτερικής πολιτικής. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Τρία λεπτά. Ο κύριος Σούλτσο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω τη σημερινή συζήτηση με εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θεωρώ πως πηγαίνει η σωστή κατεύθυνση σε αυτή στην οποία πρέπει να σκεφτόμαστε για το μέλλον, στην ανάμειξη δηλαδή των εθνικών κοινοβουλίων. Πρέπει να σταματήσουμε να θέτουμε το εθνικό εναντίον του ευρωπαϊκού. Από κοινού έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να δούμε αυτά τα οποία ε, έχουμε να κάνουμε Οπότε θα ήθελα να συμφωνήσω με τον Φιλανδό συνάδελφο που είπε πως και η πολιτική ασφάλεια πρέπει ε, να αποτελέσει αντικείμενο της υπηρεσία αυτής, η οποία θα πρέπει να είναι ανοιχτή στους ε, πολίτες. Οπότε οι προτεραιότητες πρέπει να είναι η δημοκρατία, διαφάνεια και το ζήτημα της συναπόφασης όλα αυτά πρέπει να είναι στο κέντρο της νέας υπηρεσίας. Οπότε τίθεται το ερώτημα πώς θα διαμορφωθεί το περιεχόμενο της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και εδώ πέρα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα ε, συσταθεί η νέα αυτή υπηρεσία. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ως εταίρος άλλων κρατών και περιοχών στον κόσμο, η οποία είναι υπέρ της καταπολέμησης στόχιας, υπέρ της πολιτικής επίλυσης των συγκρούσεων, υπέρ της ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. θα πρέπει να αποτελέσει το αντικείμενό μας. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ήδη από την διάρθρωση της υπηρεσίας αυτής πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει ο διάβλος που λέγεται κυρία Άστον για να διατηρήσουμε την κοινοτική ε, προσέγγιση. Εδώ πέρα συμφωνώ με τους κυρίους Μπροκ και Φερχόφστατ. Το ζήτημα είναι να διασφαλίσουμε τον έλεγχο της κοινοτικής πολιτικής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό το τονίζω και από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Χρειαζόμαστε πολύ πιο ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ Εθνικών και Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων παράδειγμα η εμπορική πολιτική, η αναπτυξιακή πολιτική. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πρέσβη, τον κύριο Κριστόφερσεν συγκεκριμένα σε περιπτώσεις συγκρούσεων πώς θα βρεθεί μία λύση χωρίς να πάνε οι κοινοτικοποιημένοι τομείς πολιτικής ξανά πίσω σε μια διακυβερνητική λειτουργία. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο κύριος Ρίτλα, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών του Κοινοβουλίου της Σλοβακίας. Για ναι, τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Θα μιλήσω γαλλικά ακολουθώντας ε, την προτροπή του Προέδρου Λαμπέρτοντίνη τη δεύτερη γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω τη λύπη μου για την απουσία της κυρίας Άστον στη συνάντησή μας αυτή. Άκουσα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την παρουσίαση την οποία έκανε ο κύριος Χριστόφερσεν. Αλλά όσο προχωράει η συζήτηση, τόσο περισσότερα προβλήματα ανακοινούνται. Και καλό θα ήταν η κυρία Άστον να μπορέσει να ακούσει από πρώτο χέρι τα προβλήματα τα οποία θέλουμε να θέσουμε. Και αν το κάνει αυτό δεν θα έχει την ανάγκη να ταξιδεύει σε 27 χώρες, γιατί θα γνωρίζει αυτά τα οποία αναμένονται από τις υπηρεσίες της. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι έχουμε μια ξεκάθαρη πολιτική βούληση από πλευράς των χωρών μελών να θέσουν σε λειτουργία την συγκεκριμένη αυτή ε, υπηρεσία. θα ήθελα να υιοθετήσω αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σιριμπέιρο Κάστρο και ο κύριος Λαμπέρτο όπως και η Γερμανίδα εκπρόσωπος. Θα ήθελα επίσης να πω στον κύριο Νταφ ότι σίγουρα η κυρία Άστον δεν μπορεί να είναι πανταχού παρούσα, αλλά θα πρέπει εν πάση περιπτώσει να μπορέσει να προγραμματίσει τα της παρουσίας της με τακτικό τρόπο, με προβλεπτό τρόπο, έτσι ώστε να ενημερώνει και να ενημερώνεται ε, για την διπλωματική της δράση. Εμείς από τη Σλοβακία εμένουμε στην σωστή γεωγραφική αντιπροσωπευτική παρουσία των κρατών μελών. Δεν θέλω να αναφερθώ σε μικρές και μεγάλες χώρες. Πολλές φορές οι μικρές χώρες στην ουσία θεωρούνται τόσο μικρές που τις αγνοούν οι μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε σχέση με αυτό. Εν πάση περιπτώσει η συγκεκριμένη αυτή πρωτοβουλία ίσως λίγο να βοηθήσει να υπάρξει λίγο περισσότερη ειρήνη στον κόσμο μας σήμερα. Καλώς. Έχουν ζητήσει άλλοι δύο το λόγο. Ένα λεπτό για τον κύριο Κάστρο για να απαντήσει στον κύριο Νταφ και ένα λεπτό στην κυρία Μουνής. Να διευκρινίσω, λέει ο κύριος Κάστρο, γιατί ίσως τελικά να μην έγινε απόλυτα κατανοητός. Εγώ δεν είπα ότι η κυρία Άστον είναι υποχρεωμένη να ε, παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ λέγω ότι ε, τη συμβουλεύω να το κάνει και στα εθνικά κοινοβούλια. Δεύτερον, δεν είναι απαραίτητο να πάει μόνη της ε, ή να πηγαίνει η ίδια, εν πάση περιπτώσει, να συζητήσουν ε, με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές διάφορα θέματα. Αυτό μπορεί να γίνει και από άλλα στελέχη της υπηρεσίας της. Θα προτιμούσα βέβαια η κυρία Άστον να ήταν παρούσα εδώ σήμερα. Ευχαριστώ κύριε Βιμπέρο Κάστρο. Εγώ όμως θα σας μιλήσω στα ισπανικά, που θα είναι μια γλώσσα εργασία για την υπηρεσία τη εξωτερική δράση. Εγώ μια ομάδα εργασία για την πρόληψη των, των συγκρούσεων και κρίσεων και λέει το άρθρο 3 των προτάσεων αυτών λέει ότι ο προγραμματισμός όσον αφορά την αντίδραση σε κάποιες κρίσεις όπως ε, ορίζονται στο άρθρο 3 αυτού του, του όργανου σταθερότητας είναι κάτι το οποίο θα το αναλάβει η εξωτερική υπηρεσία. Όμως αυτή η ομάδα του προγραμματισμού της, ε, της RELEX 2 δεν προβλέπεται ε, να υπαχθεί στην νέα υπηρεσία. Επομένως ε, αυτή η αρμοδιότητα θα πάει στο Συμβούλιο και άρα έτσι θα καλυφθεί η πτυχή ασφάλεια. Επομένως, η δεύτερη ομάδα της Relax, όπως σήμερα λειτουργεί, θα έπρεπε να υπαχθεί στην νέα υπηρεσία. Δεν θα έπρεπε να υπαχθούν ε, ε, αυτές οι υπηρεσίες στο Συμβουλίο. Θα έπρεπε να καινούργια υπηρεσία. Επίσης, αυτό το ψήφισμα της 21ης πέμπτου του, του, του Γαλλικού Κοινοβουλίου λέει ότι δεν υπάρχει καμία αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λέει η Γαλλική Εθνοσυνέλευση η Γερουσία, ούτω ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφαίνεται επί τη ε, της νέα αυτή υπηρεσία. Πάρα πολύ με ξενίζει αυτό το ψήφισμα. Bene. Ε, Μετά από την τελευταία αυτή παρέμβαση θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Κριστόφερσεν. Αν μπορεί παρακαλώ να μην ξεπεράσει τα 10 λεπτά. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο αυτό. Αλλά υπήρξαν κάποιες ερωτήσεις βέβαια, υπήρξαν όμως και πολλά σχόλια. Αν μπορεί παρακαλώ να δώσει απαντήσεις στις συγκεκριμένες ερωτήσεις και τα σχόλια θα βρουν τη θέση τους στα πρακτικά της συνάντησης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις σας και για τα σχόλιά σας βέβαια. Νομίζω ότι χωρίς να μπορώ να ερμηνεύσω πλήρως αυτά τα οποία είπαν ε, οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων, μπορώ να διακρίνω νομίζω μία βασική υποστήριξη. Κάποια από τα σχόλια αφορούν τις σχέσεις μας ε, με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε εδώ να σας θυμίσω ότι ήταν στη συνάντηση τον Φεβρουάριο των Προέδρων των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπεσχέθη τότε η κυρία Άστον ότι θα συμμετέχει ε, κάθε ε, έξι μήνες στην συγκεκριμένη συνάντηση, τακτική συνάντηση. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα απλά. Όπως είπα, θα ήθελε να είναι παρούσα εδώ σήμερα, αλλά ε, συμμετέχει σε μια συνάντηση κορυφής και δεν είναι δυνατόν να είναι όπως είπαμε πανταχού παρούσα. Το θέμα των υπαλλήλων. Και σε ποιο βαθμό θα είναι στην διάθεση και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια υπηρεσία η οποία θα έχει σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτό είναι μέσα στις αρμοδιότητές μας. Και δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία διαφοροποίηση σε σχέση με αυτή τη διαπίστωση. Η υπηρεσία αυτή θα ενημερώνει ε, αν θέλετε, σε τακτική ή όχι βάση και τα εθνικά κοινοβούλια με τον ίδιο τρόπο που θα ενημερώνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε περισσότερη διαφάνεια και ε, να έχουμε καλύτερη κατανόηση της δράσης μας. Τα κοινοβούλια των χωρών μελών έχουν ένα σαφέστατο πολιτικό ρόλο να παίξουν γύρω από τον καθορισμό των έπαιξαν και όλα σε ένα συγκεκριμένο ρόλο σε σχέση με τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων α, της υπηρεσίας μας στα πλαίσια της, εξω, της ΚΕΠΑ, της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας που εντάσσεται στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου και των α, Κοινοβουλίων. Τέθηκαν αρκετές ερωτήσεις για το πόσο φιλόδοξη είναι η υπηρεσία αυτή ή πόσο φιλόδοξη θα πρέπει να είναι η υπηρεσία αυτή. Ο κύριος Ντίνη είπε ότι υπάρχουν κάποια όρια προς την κατεύθυνση αυτή. Αν θέλει κανείς να συμπεριλάβει όλους τους τομείς πολιτικής που έχουν και κάποιες εξωτερικές πλευρές, τότε στην ουσία θα πρέπει να εντάξει στην υπηρεσία αυτή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί πιστεύουν σαν παράδειγμα ότι η ενεργειακή πολιτική σε σχέση με την προμήθεια ενέργειας, σε σχέση με τη μόλυνση, σε σχέση ε, με την ε, συνέπειες των κλιματολογικών αλλαγών, όλα αυτά θα μπορούσαμε να τα επιδιώξουμε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε κάπως επιφυλακτικοί. Και η πρόταση την οποία ουσιαστικά κάνουμε είναι μια υπηρεσία η οποία να συμπεριλαμβάνει κάποιες από τις σημαντικές πλευρές της αναπτυξιακής πολιτικής παρότι θα υπάρχει όπως είπα ένας ανεξάρτητος επίτροπος για τα θέματα αυτά στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και η υπηρεσία μας αυτό το οποίο θα προσπαθεί να κάνει είναι να εξυπηρετεί τον αρμόδιο επίτροπο και για τα θέματα της πολιτικής γειτονίας. Εκεί θα λειτουργεί η εξωτερική αυτή η υπηρεσία, θα έλεγα σχεδόν κατά αποκλειστικότητα. Πάντως η υπηρεσία αυτή δεν είναι, επαναλαμβάνω, μια υπηρεσία για την κυρία Άστον. Είναι μια υπηρεσία η οποία θα είναι στη διάθεση του συνόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλων των άλλων οργάνων μεταξύ του οποίων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ας πάρουμε το παράδειγμα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αν δει κανεί την κατάσταση στην Αϊτή, έχουμε να κάνουμε με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας έκτακτη κατάστασης τα μέσα τα οποία υπάρχουν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο εσωτερικό της νέας αυτής υπηρεσίας τέθηκαν στη διάθεση της ευρωπαϊκής δράσης και παρουσία στην ΑΕΤ. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι απαραίτητο να εντάξουμε το σύνολο της υπηρεσίας ΕΚΟ στα πλαίσια της εξωτερικής αυτής νέας υπηρεσίας. Για κάποιες περιπτώσεις Ίσως ε, για πολιτικούς λόγους ή για πρακτικούς λόγους θα είναι ένα πλεονέκτημα η συμπερίληψη της ΕΚΟ στις δραστηριότητες της εξωτερικής υπηρεσία, ίσως και όχι. Τώρα για την στρατιωτική δομή. Νομίζω ότι αυτά τα οποία έχουμε οικοδομήσει ε, τα τελευταία χρόνια είναι κάποιες ικανότητες στρατιωτικές και πολιτικές στο εσωτερικό της υπηρεσίας αυτής, της, της υπηρεσίας του Συμβουλίου καταρχάς, που θα ενταχθούν τώρα στις ε, δυνατότητες και τις ικανότητες που θα έχει η νέα υπηρεσία. Είναι ένα πλεονέκτημα. Λίγοι έχουν αυτό το πλεονέκτημα στον κόσμο. Αυτός ο συνδυασμός στρατιωτικής και πολιτικής δράσης, όπως είδαμε να λειτουργεί τα τελευταία χρόνια, έχει συνεισφέρει τα μάλα στην εφαρμογή των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, σαν παράδειγμα, σε αρκετά μέρη του κόσμου. Υπήρξαν και αρκετές ερωτήσεις σχετικά με το κόστος. Το πρώτο σχόλιο το οποίο θα ήθελα εδώ να κάνω γύρω από θέματα κόστους είναι ότι σήμερα Υπάρχουν στα πλαίσια των δυνατοτήτων της εξωτερικής πολιτικής κάποια, κάποια τμήματα του προσωπικού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη Γραμματεία του Συμβουλίου. Όπως επίσης και στα πλαίσια της Γραμματείας της Εναλλασσομένης Προεδρίας, όλοι αυτοί ασχολούνται με την εξωτερική πολιτική. και ακόμα και οι μόνιμες αντιπροσωπείες της Βρυξέλλες όταν αναλαμβάνει η χώρα τους μια προεδρία αν ενισχύουν το προσωπικό τους και συμπληρώνονται. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε απλά να συνδυάσουμε με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο όλα τα μέσα και τις δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό θα είναι το δύσκολο. Δεν υπάρχει αμφιβολία λοιπόν τώρα που θα αναλάβουμε όλες αυτές τις υπηρεσίες. Τώρα που θα είναι υπεύθυνη η εξωτερική υπηρεσία για τον συντονισμό όλων αυτών των ομάδων, ότι θα απαιτηθεί επιπλέον προσωπικό. Αυτό δεν είναι έκπληξη για κανένα. Και αυτό σημαίνει φυσικά επιπλέον κόστος. σε ένα βαθμό το κοινοτικό προσωπικό θα αντικαταστήσει το εθνικό προσωπικό το οποίο λειτουργούσε προσωρινά θα έλεγα σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια των προεδριών κτλ. Αυτό το επιπλέον προσωπικό θα είναι ένα από τα μέσα με τα οποία θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ε, το αργότερο το 2013 η υπηρεσία να αποτελείται ε, κατά το 1 τρίτο τουλάχιστον στην κατηγορία προσωπικού α από ε, στελέχη τα οποία θα προέρχονται από τα κράτη-μέλη. Κάποια στελέχη θα έρθουν απευθείας από τα κράτη-μέλη. Ε, κάποιοι εμπειρογνώμονες εθνικοί θα μπορεί να μετατραπούν σε εισαγωγικά σε θέσεις υπαλλήλων α. Τέθηκε το θέμα πόσο χρόνια θα παραμένουν στις θέσεις αυτές οι εθνικοί διπλωμάτες. Εμείς είπαμε ότι αυτό μπορεί να μένει μέχρι 10 χρόνια. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω θα έλεγα και να συζητηθεί όταν ξεκινήσει και η λειτουργία αυτής της υπηρεσίας. γιατί δεν νομίζω ότι θα είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής όταν η υπηρεσία θα μπορούσε να αποτελείται αποκλειστικά από προσωπικό το οποίο θα εναλλάσσεται σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Αυτά θα τα δούμε όμως και το 2013. Ο κύριος Ντίνη αναφέρθηκε στα θέματα των ευθυνών και το σε ποιον θα είναι υπόλογη η συγκεκριμένη υπηρεσία. Για το θα υπάρχει δηλαδή δημοκρατικό έλεγχο, οπότε σε αυτή την περίπτωση όλα αυτά θα πρέπει να ενσωματωθούν σε κάποια κείμενα νομικά δεσμευτικά, θα ενταχθούν και αυτά στη διοργανική συμφωνία ή θα μπορούν να περάσουν και από αναθεώρηση και κατά αυτόν τον τρόπο θα κατοχυρωθούν τα όσα προβλέπονται. Επίσης, επιτρέψτε να προσθέσω τα εξή. Για τις θετικές τη συνεργασία ε, συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτή που έλαβε χώρα τον ε, περασμένο μήνα, είναι το ότι στην τελική μας απόφαση θα προβλέπεται ε, ο έλεγχο του προπολογισμού, θα προβλέπεται απαλλαγή όσον αφορά τον προπολογισμό. Επομένω, κάνουμε ό,τι μπορούμε τόσο ώστε να εξασφαλίσουμε πω θα υπάρχει όσο γίνεται περισσότερη διαφάνεια όσοι γίνεται και ότι θα υπαγόμαστε και εμεί στην διαδικασία του ελέγχου του προπολογισμού ε, στην απαλλαγή. Ό,τι ισχύει ακριβώ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα. Ε, ελπίζω ότι απάντησα όσο, όσο γίνεται περισσότερο. Σα ευχαριστώ που δεχτήκατε να κλείσετε. Προφανώς δεν έχουμε καλύψει όλα τα θέματα, αλλά πρέπει να σεβαστούμε, θα έλεγα, με οικονομικό τρόπο τον χρόνο τον οποίο έχουμε μπροστά μας. Ίσως ε, δεν πήραν όλοι όσοι θα επιθυμούσαν τον λόγο. Διατηρώ τον κατάλογο αυτό για την επόμενη συζήτηση, αλλά θα ήθελα να δώσω το λόγο για να σεβαστούμε την ημερήσια διάταξή μας στην αρμόδια υπάλληλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θα παρουσιάσει το νομικό πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής μέσα στο επόμενο δεκάλεπτο. Okay, so thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ανέφερε και ο κύριος Κριστόφερσεν, η σύσταση αυτής της υπηρεσίας απαιτεί κάποια νομοθετικά μέτρα, ένα από τα οποία είναι η τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και λοιπόν υπαλλήλων. Αυτό θα γίνει υπό την τακτική νομοθετική διαδικασία, δηλαδή θα αναμειχθεί πλήρως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρώτα απ' όλα, πριν περάσουν ουσία, να σας ενημερώσω λίγο στο... για το πού βρισκόμαστε όσον αφορά την πρόταση της Κομισιόν. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις με τα συνδικάτα και συζητάμε τώρα το κείμενο στην Επιτροπή Κανονισμού που συμπεριλαμβάνει εκπροσώπους ε, των διοικήσεων και των συνδικάτων από όλα τα θεσμικά όργανα, η οποία πρέπει να γομοδοτήσει μέχρι αύριο και η Κομισιόν αναμένει να υιοθετήσει την επίσημη πρότασή της την ερχόμενη εβδομάδα στις 9 Ιουνίου και μετά βέβαια θα ακολουθήσει η κανονική διαδικασία διαβούλευσης, υποβολή δηλαδή της πρότασης στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω πως ο κανονισμός αυτός αποτελεί το βασικό πλαίσιο εντός του οποίου ε, θα γίνει η πολιτική προσωπικού της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Αυτό σημαίνει πως ο ύπατος εκπρόσωπος θα πρέπει να η είπατε εκπρόσωπος θα πρέπει να προχωρήσει σε κάποιες εφαρμοστικές διατάξεις για να περάσουμε στην επιχειρησιακή φάση. Όταν μιλάμε λοιπόν για την ουσία των προτινόμενων αλλαγών, το σημαντικό είναι το άρθρο 27 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με αυτό το άρθρο, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα συμπεριλαμβάνει υπαλλήλου που θα προέρχονται από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, την Κομισιόν και προσωπικό αποσπασμένο από τις Εθνικές Διπλωματικές Υπηρεσίες των Κρατών Μελών. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε πως το προσωπικό από αυτές τις τρεις πηγές θα έχει την ίδια ακριβώς αντιμετώπιση. Αυτό σημαίνει πως όταν θα τροποποιήσουμε τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης θα πρέπει να διασφαλίσουμε πως οι υπάλληλοι Συμβουλίου Κομισιών και οι εθνικοί διπλωμάτες θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Οπότε δεν θα δίνεται προτεραιότητα σε εσωτερικούς φωσφίους όταν ε, προκυρήσονται θέσεις. Επίσης, για να υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση από τις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες, θα μπορούμε μέχρι την 30 Ιουνίου 2013, δηλαδή αυτό το οποίο λέμε την αρχική φάση, να λάβουμε ιδιαίτερα μέτρα για να διευκολυνθεί η ενσωμάτωσή τους, κάτι το οποίο σημαίνει πως στην περίπτωση στην οποία έχουμε ανοιχτές θέσεις. Εάν χρειάζεται να ενσωματώσουμε αυτούς τους υπαλλήλους, θα τους δοθεί προτεραιότητα ε, σε περίπτωση που μιλάμε για ανθρώπους με παρόμοια προσόντα. Μετά από αυτή την αρχική φάση που θα τελειώσει 30 Ιουνίου 2013 θα υπάρχει ίση πρόσβαση και σε υπαλλήλους από άλλα θεσμικά όργανα. Θα ήθελα τώρα να μείνουμε στο ζήτημα των ατόμων που θα προέρχονται από τις εθνικές διπλωματικές αρχές. Για να ενσωματωθούν στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης δημιουργούμε μια ιδιαίτερη κατηγορία συμβασιούχων, θα λέγαμε, η οποία θα ομοιάζει στο μέτρο του δυνατού αυτή των υπαλλήλων. Δηλαδή θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις η διάρκεια των συμβασιών τους προβλέπεται να είναι μια αρχική περίοδο τεσσάρων ετών που θα μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για τέσσερα έτη υπό την προϋπόθεση βεβαίως πως τα κράτη-μέλη από τα οποία προέρχονται θα συμφωνούν. Την πρώτη ημέρα, όπως ορίζει η απόφαση του Συμβουλίου, κάποιες οντότητες Συμβουλίου και Κομισιόν θα μεταφερθούν στην υπηρεσία αυτή, οπότε και το προσωπικό που τις αποτελεί. Επιπλέον. Για τους υπαλλήλους που θα μεταταγούν σε αυτή την υπηρεσία, εάν θέλουν να επανέλθουν στο θεσμικό όργανο από το οποίο προήλθαν, θα έχουν προτιμησιακή μεταχείριση έτσι ώστε να μπορούν να ε, ζητήσουν θέσεις οι οποίες ανοίγουν στο ίδιο πέδο με τους εσωτερικούς υποψηφίους. Θα ήθελα τώρα να σας πω κάποια πράγματα περισσότερο για την συγκεκριμένη κατάσταση των αντιπροσωπιών. Και μετά θα μιλήσουμε για τους επικεφαλείς των αντιπροσωπιών και μετά για τις ελέγχου των αντιπροσωπιών. Οι επικεφαλείς των αντιπροσωπιών. Η Κομισιόν θα αναμειχθεί στον ορισμό τους, στο μέτρο κατά το οποίο μπορούν να διοριστούν με βάση μια λίστα προεπιλογής ε, στην οποία θα έχει συμφωνήσει η Κομισιόν. Όσον αφορά τις αντιπροσωπείες της Ένωσης, σε αυτές τις αντιπροσωπείες όπως ξέρετε θα έχουμε προσωπικό της Κομισιόν το οποίο θα συνυπάρχει με προσωπικό της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Αυτό σημαίνει πως όσον αφορά θέματα διοικητικά, οργανωτικά και οικονομικά θα λαμβάνουν οδηγίες οι υπάλληλοι της Κομισιόν από τον επικεφαλής αντιπροσωπείας, ο οποίος ανήκει στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Από την άλλη, η υπηρεσία, το προσωπικό της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, το οποίο θα διεξάγει καθήκοντα της Κομισιόν, θα λαμβάνει οδηγίες από την Κομισιόν επ' αυτών. Επιπλέον, υπάρχουν και κάποιες άλλες τεχνικές ε, τροποποιήσεις με τις οποίες δεν θα σας απασχολήσω και νομίζω θα μείνω σε αυτά για να έχουμε χρόνο για συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κυρία Σούκα για την παρουσίασή της. Όπως είπα, έχω 12 εγγεγραμμένους ομιλητές. Πρώτος ο κύριος Γκουαλτιέρη, εισηγητής της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων που είναι υπεύθυνη και για τον κανονισμό των υπαλλήλων. Τέσσερα λεπτά. Ελπίζω να μπορέσεις να σεβαστείς το τετράλεπτο. Ευχαριστώ. Εγώ εκπροσωπώ εδώ τον εισηγητή, τον Ράπκε, ο οποίος μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω. Θα ήθελα να πω ότι ο κανονισμός για το προσωπικό είναι ένα σημαντικό θα έλεγα στοιχείο της δημιουργίας της νέας υπηρεσίας. Θα έλεγα δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί αυτό και ο καθορισμός των τρόπων με τους οποίους θα λειτουργεί η υπηρεσία αυτή ε, είναι κάτι το αρκετά σημαντικό, για να μην πω το κομβικό σημείο του τρόπου λειτουργίας ε, της συγκεκριμένης υπηρεσίας και γι' αυτό ακριβώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περίμενε ε, πριν περάσει στην συγκεκριμένη υιοθέτηση αυτής της πρότασης την επίσημη πρόταση τροποποίησης του κανονισμού των υπαλλήλων. Όπως και να έχουν τα πράγματα, οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι γνωστές, έχουν επαναληφθεί σε πολλές συναντήσεις της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Ξεκινώντας θα έλεγα από μια μεθοδολογική προκαταρκική παρατήρηση. Λέμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η νομική βάση η οποία είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί για την μεταρρύθμιση του κανονισμού έτσι όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο άρθρο 37 ορίζει ότι ουσιαστικά η, το άρθρο 6 της απόφασης του Συμβουλίου δεν μπορεί να ορίσει σε λεπτομερές επίπεδο τους τρόπους με τους οποίους θα γίνει η μεταρρύθμιση της υπηρεσίας αυτής. Οι αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν σύμφωνα με την διαδικασία της συναπόφασης. Γίνεται μια προσπάθεια από πλευράς ε, του κυρίου Κριστόφερσεν και της υπηρεσίας του, έτσι ώστε να βελτιωθεί η διατύπωση του άρθρου 6 διευκρινίζοντας ότι τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνει το άρθρο 6 είναι ε, αρχές ουσιαστικά οι οποίες δεν φύγουν και δεν είναι αντίθετες με τις κοινοτικές διαδικασίες. Είναι σαφές ότι οι συγκεκριμένες αυτές διατυπώσεις μπορούν και να βελτιωθούν αλλά σίγουρα συνιστούν ένα σημαντικό πρώτο για να έλθω τώρα στην ουσία των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ισοτιμία αντιμετώπισης καθηκόντων και υποχρεώσεων και δικαιωμάτων έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν σαν ένα πραγματικά ευρωπαϊκό σώμα. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες γίνονται. Η πρώτη αφορά το ότι αυτοί οι εθνικοί εμπειρογνώμονες, ε, οι αποσπασμένοι, δεν θα πρέπει να δημιουργήσουν, αν θέλετε, αυτό που θα ονομάζαμε μια τέταρτη κατηγορία και θα πρέπει ο αριθμός τους να ελέγχεται κάθε φορά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι οι συμβασιούχοι οι οποίοι θα προέρχονται από τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να παραμένουν στην υπηρεσία και τέλος υπάρχει και το επίσης σημαντικό θέμα που αφορά τις ποσοστώσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει ξεκαθαριστεί ότι το 1 τρίτο θα πρέπει να προέρχεται από τα κράτη-μέλη. Είναι σαφές όμως ότι τουλάχιστον το 50% θα πρέπει να προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί το ποσοστό των κοινοτικών αρμοδιοτήτων που έχει η υπηρεσία αυτή ε, το καλεί αυτό θα έλεγα, το απαιτεί. Ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρξει και ισορροπία ε, γεωγραφική θα έλεγα, κάτι το οποίο συνηθίζεται και νομίζουμε επίσης ότι και η ετήσια έκθεση ε, της του εκπροσώπου ε, θα πρέπει να παρουσιάζεται, να κατατίθεται και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Γκαλτιέρη. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Πορτογαλικής Βουλής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω και εγώ κάποια σχόλια τα οποία θα ήθελα να κάνω και κάποιες ερωτήσεις που επικεντρώνονται σε δύο στοιχεία. Πρώτα απ' όλα τα κριτήρια για τον ορισμό διπλωματών και υπαλλήλων. Δεύτερον, η ανάγκη να αποφευχθούν συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Νομίζω πως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα κριτήρια ορισμού όπως ε, σας είπα, να ληφθούν δηλαδή υπόψη και ιστορικοί δεσμοί και γεωγραφική εκπροσώπηση. Ε, ιστορικοί δεσμοί οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο και όσον αφορά τις γλώσσες. Θα ήθελα να ακούσω κάτι από αυτό. Νομίζω πως αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς πρέπει να ενισχύσουμε την παρουσία και το προφίλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ταυτόχρονα όμως αυτό δεν σημαίνει η αποδυνάμωση των ε, κρατών μελών στις ε, εξωτερικές τους ε, πολιτικές. Ένα άλλο στοιχείο που μας ανησυχεί αφορά την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να αποδεικτούν αυτές οι συγκρούσεις γιατί ανησυχώ. Έχουμε ήδη δει έναν βαθμό ανταγωνισμού μεταξύ ε, Συμβουλίου και Κομισιών και φοβάμαι πως αυτό μπορεί να μεταφερθεί στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης και να καταλήξουμε σε έναν ανταγωνισμό μεταξύ της υπηρεσίας αυτής και των κρατών μελών, παρά το ότι ε, προβλέπεται η σχέση τους να είναι συμπληρωματική. Αν μπορείτε λοιπόν να σχολιάσετε αυτά τα δύο, Ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπος τώρα της Γαλλικής Γερουσίας για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα να σας πω, κύριε Πρόεδρε, αφορά το, το, ε, αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος, ο οποίος με κάλυψε και γιατί έχει εργαστεί πάνω στα θέματα αυτά στην ε, Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Θεμάτων και τελευταίες 15, 15 ε, μέρες αλλά και εβδομάδες και χρόνια θεωρούμε ότι ε, θα πρέπει να προβάλλεται περισσότερο η διαδρομή για το έργο της Ευρώπης ε, θα πρέπει να μετράει περισσότερο η Ευρώπη όσον την επίλυση των διεθνών κρίσεων. Μέση Ανατολή, Ασία, υπερθερμές του πλανήτη, το πυρηνικό πρόβλημα με το Ιράν δεν μπόρεσε τελικά να είναι καταλήτης εξελίξεων η Ευρώπη. Δεν έχει την αξιοπιστία που πρέπει και για να την αποκτήσει πρέπει να μιλά με μία φωνή στη διεθνή σκηνή. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε παρά να είμαστε υπέρ του να συγκροτηθεί μια τέτοια υπηρεσία εξωτερική δράση. Τώρα, θα ήθελα να επανέλθω στο εξή. Βεβαίω, είναι απαραίτητο να υπάρχει μια εξωτερική πολιτική, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε το ότι για μας οι αποφάσεις που μας δεσμεύουν για στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά επίσης όσον αφορά και τη δημοσιονομική κάλυψη της υπηρεσίας, είναι για μας κάτι που θα πρέπει να ρυθμίζεται σε διακυβερνητικό επίπεδο και να ελέγχεται από τα εθνικά κοινοβούλια. Όχι, δεν θέλουμε να γίνεται η υποστήριξη αυτών των επιχειρήσεων από τον κοινωνικό προπολισμό, όπως ας πούμε για το Αφγανιστάν. Ακριβώς αυτό ίσχυσε εκεί. Πολλές φορές μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά τα οποία χρειάζεται να εκταμιεύονται. Αυτά. Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Μπουλά. Συνάδελφος Σάριος Βόλσκι. για την τροποποίηση του κανονισμού του υπαλληλικού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα να συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπε ο κ. Κριστόφερσον όσον αφορά την προσέγγιση των θέσεων μας. Αυτό είναι εμφανές. Πάντως έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας και δουλειά να κάνουμε. Έχουμε το έγγραφο Verhofstadt Μπροκ, όπου διατυπώνει τη θέση του Κοινοβουλίου και στις σχετικές τροπολογίες. Αυτές που ε, αποσκοπούν στο να τροποποιήσουν την ε, απόφαση του Συμβουλίου και είπαμε ότι θέλουμε εμείς και η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο μας ισχυρή τέτοια υπηρεσία ε, να έχει βεβαίως την δημοκρατική νομιμότητα που απαιτείται και επομένως να είναι υπόλογη στον κοινωνικό έλεγχο τώρα. Για το προσωπικό είχαμε τα, τις προτάσεις του Γενικού Διευθυντού. Θεωρώ ότι επιδέχεται βελτιώσεις, επιδέχεται περισσότερη προσέγγιση θέση ε, όπως παρουσιάστηκε αυτή με τις θέσεις του Κοινοβουλίου. Γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα, αυτό θέλουμε, στην ε, νέα υπηρεσία. όλα τα κράτη-μέλη, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αισθάνεται δική τη την υπηρεσία, τόσο ώστε να μπορεί να ταυτίζεται με τι ενέργειε τη υπηρεσία αυτή από την πρώτη μέρα λειτουργία τη. Θα πρέπει να έχουμε ε, φυσικά αξιοκρατία, αλλά αξιοκρατία που να συνδυάζεται με γεωγραφική εκπροσώπηση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, βέβαια και η εμπειρογνωμοσύνη δεν είναι ουδέτερη γεωγραφικά. Εκπαίδευση διπλωματών, ε, και βέβαια για να είναι άρτη αυτή η εκπαίδευση θα πρέπει οι εκπαιδευτέ να προέρχονται από όλη την Ευρώπη. Να ληφθεί υπόψη το άρθρο 87 του κανονισμού και η Ρέλεξ που θα είναι η πηγή από την οποία θα ξεπηδήσει μια υπηρεσία ε, δεν είναι εκεί πάρα πολύ ευέλικτη. Μάλτα 0%, Βουλγαρία 16%, Κύπρος 16% και το Λουξεμβούργο 18%, η Ρουμανία 18% και η Λετωνία 20%, Πολωνία 26%, Σλοβενία 28%, 33 ε, Λιθουανία, Στονία 33, Τσεχία 344, η Γερμανία 70%, σε 73 η Βρετανία και 95 η Ιταλία. Μα γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν χρησιμοποιεί ε, τον σχετικό κανονισμό ούτως ώστε να έχει κάποιο νομικά δεσμευτικό νομοθέτημα ούτως ώστε να υπάρχει ε, μια, μια, μια αντιπροσωπευτικότητα που θεωρητικά την αποδέχεται. Ευχαριστούμε κύριε Σάλους Βόλτς κύριε πρόεδρος. Και τώρα το λόγο για κύριο Σεβερίν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να κάνω κάποιες πιο γενικές ε, παρατηρήσεις. Είναι προφανές πως μιλάμε για ένα τεχνικό ε. μέσο και όχι για μια πολιτική απόφαση. Οπότε από αυτή τη σκοπιά πρέπει να αντιληφθούμε πως το μέσο αυτό είναι και πρέπει να είναι θετικά νέα για τους πολίτες μας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί συνεχώς μας ζητάνε μέσω διαφόρων δημοσκοπήσεων πως θέλουν περισσότερη αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, συνεκτικότητα στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Αυτό είναι επίσης καλά νέα για τους συνομιλητές μας, ε, παγκόσμιους παίκτες όπως είπα Κίνα, Ρωσία που ζητάνε συνεχώς μεγαλύτερη συνεκτικότητα και σαφήνεια στις σχέσεις ε, με αυτούς. Οπότε δεν είναι θέμα νέων αρμοδιοτήτων προς το Κοινοβούλιο ή την Κομισιόν, αλλά είναι καλό να έχουμε ένα πιο αποτελεσματικό μέσο στη διάθεσή μας ταυτόχρονα. Θεωρώ πως δεν πρέπει να είναι ακριβώς ε, μόνο αποτελεσματικό τεχνικά το μέσο αυτό, αλλά και ευρωπαϊκό. Οπότε το θέμα δεν είναι η αντιπροσωπευτικότητα, αλλά η ικανότητα να εκπληρώσει μια αποστολή. Η γεωγραφική ισορροπία όμως σημαίνει ισορροπία ευαισθησιών και γνώσεων και βεβαίω δεν είναι θέμα αντιπροσωπευτικότητας αλλά ισορροπίας δυνατοτήτων ή να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις για τα εθνικά κοινοβούλια οπωσδήποτε θα συνεχίσουν να έχουν τις ίδιες δυνατότητες ελέγχου των κυβερνήσεών τους μέσω του Συμβουλίου και βεβαίως την δυνατότητα να συνομιλούν μαζί μας και να συνεργάζονται μαζί μας. Οπότε αυτό το οποίο θα πω τελευταίο είναι πως για το προσωπικό πρέπει να φροντίσουμε πως το προσωπικό θα είναι πιστό, εάν θέλετε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι προς τις χώρες προέλευσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σεβερίν. Ο κύριος Τεμπεστίνη από την Ιταλική Βουλή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η απουσία της κυρίας Άστον είναι κάτι το οποίο με δυσαρεστεί. Βέβαια αυτό το οποίο έχει σημασία κατά τη διάρκεια των επομένων μηνών να μπορέσουμε να ακαλύψουμε τις καθυστερήσεις τις οποίες έχουμε σημειώσει όπως υπογράμμισαν και οι Γάλλοι συνάδελφοι στον τομέα της ΚΕΠΑ. Θα ήθελα να καταλήξουμε το ταχύτερο δυνατόν σε μια κάποια συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό ακριβώς και υποστηρίζουμε τις απόψεις και του κύριου Φερχόφστατ και του κύριου Μπρόκ. Έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, η οποία ξέρουμε πώς δημιουργήθηκε, έχει θα έλεγα διακυβερνητική προέλευση, να μην λειτουργήσει σαν μια τροχοπέδη στην εξέλιξη των εξωτερικών πολιτικών, αλλά να βοηθήσει το κοινοτικό θα έλεγα πρόγραμμα. Θα ήταν πράγματι ε, μεγάλο λάθος μια τέτοια υπηρεσία να ενσωματώσει ε, κάποιες λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να μεταφέρει τις υπηρεσίες αυτές, όπως έλεγε ο κ. Φερχόφστατ, από το κοινοτικό στο διακυβερνητικό επίπεδο. Αντίθετα, η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να αποτελέσει ένα βήμα προς τα εμπρός στα πλαίσια της κοινοτικής ολοκλήρωσης. Είναι προφανές ότι οι εθνικές διοικήσεις ζητούν και το κοινό γενικότερα ζητά ε, μια Ευρώπη περισσότερο διαφανή, μια Ευρώπη η οποία να ασκεί μια κατανοητή εξωτερική πολιτική. Και εδώ ακριβώς έρχεται και το θέμα της σχέσης με τα Εθνικά Κοινοβούλια και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε μαζί με την υπηρεσία αυτή και η ΜΕΝ και η ΔΕ και η συγκεκριμένη υπηρεσία θα πρέπει να μάθει να βρίσκει τους σωστούς συνομιλητές και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε επίπεδο Εθνικών Κοινοβουλίων έτσι ώστε η εξωτερική αυτή υπηρεσία να φέρει πέρα στην αποστολή της σωστά. Ευχαριστώ κύριε Τεμπεστίνη. Εκπρόσωπος του Bundestag. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα έχω κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα για το προσωπικό. Θα ήθελα να γνωρίζω τι γίνεται με το δικαίωμα επιστροφής ε, συνεργατών που προέρχονται από τα κράτη-μέλη. Αν θέλουν να επιστρέψουν δηλαδή στα κράτη-μέλη τους, τι ε, πρόβλεψη υπάρχει, εάν υπάρχει. Δεύτερο συγκεκριμένο ερώτημα αναφέρεται στον ε, κατάλογο της ε, είπα της Εάν ε, δεν συμφωνεί η Κομισιόν σημαίνει αυτό πως έχει μετά δικαίωμα βέτο και μια τελευταία ερώτηση Να πω γιατί ε, φαίνεται πως ακούσαμε κάποια πράγματα τα οποία οφείλονται σε άγνοια αφενός για τις στρατιωτικές αποστολές ε, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό δεν ψηφίζονται πλέον από την Βουλή, όπως και οι εκπαιδευτικές αποστολές. Στη Σομαλία δεν ψηφίσαμε καθόλου και εκεί πέρα δεν υπήρχε καμία συμμετοχή της Γερμανικής Βουλής. Θέλω να ξεκαθαρίσω για όσους δεν γνωρίζουν πάρα πολύ τα, του γερμανικού δικαίου και των δικαιωμάτων της Γερμανικής Βουλής. Κατόπιν, να αναφέρω πως πάρα πολλοί οργανώσεις αναπτυξιακής βοηθείας, γαλλικές, γερμανικές, αγγλικές, ε, αλλά νομίζω αυτό μπορούν να το βεβαιώσουν και οι πράσινοι και οι σοσιαλδημοκράτες συναδελφοί και θα τους ενδιαφέρει, ε, είναι πως αυτές οι οργανώσεις ασκούν κριτική ή κάνουν ερωτήματα για το εάν η υπηρεσία αυτή όπως έχει μέχρι τώρα όπως φαίνεται ότι θα οργανωθεί, εάν είναι σύμφωνη με την συνθήκη. Υπάρχουν πάρα πολλές νομικές γνωμοδοτήσεις από πάρα πολλά δικηγορικά γραφεία που έλαβαν εντολή από αυτές οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και κατέληξαν πως ε, από μια γενική υπηρεσία εκπροσώπηση, δεν γίνεται λόγος μάλλον για κάποια ε, υπηρεσία γενικής εκπροσώπησης στη συνθήκη της Λισαβόνας, οπότε δεν ξέρουν κατά πόσον στέκει όπως έχει συσταθεί η υπηρεσία εξωτερικής ε, δράσης και αυτό συνδέεται βεβαίω με την κριτική του ότι υπάρχει συνεχώς μία σύνδεση ε, πολιτικής και στρατιωτικής πτυχής, καθώς φαίνεται πως ε, η πολιτική πτυχή θεωρείται μάλλον συμπλήρωμα και όχι εναλλακτική λύση στην στρατιωτική δράση. Οπότε θα ήθελα εδώ πέρα να ζητήσω από τους συναδέλφους να σκεφτούν αυτή την κριτική και τις αμφιβολίες ακριβώς τώρα που μιλάμε για τη σύσταση της υπηρεσίας αυτής και τέλος να απευθυνθώ στον κύριο Ντίνη και να τον υποστηρίξω σε αυτά τα οποία είπε πως πρέπει να είναι σαφές πως οι στρατιωτικές ε, αυτές αποστολές πρέπει να ελέγχονται. Σας ευχαριστώ. Αούταλα τώρα πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε πρόεδρε. θα θέλω να σας τονίσω. Θα σας τονίσω το πόσο σημαντική είναι η πολιτική για την πρόσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε εδώ τα Εθνικά Κοινοβούλια γιατί πολλές φορές τα ξεχνάμε αυτά. Ακόμα και αν αποτελούν θεμέλιο λίθο όπως και η δημοκρατία βέβαια για την, ε, για την Ευρώπη. Επομένως, όλοι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι καινούργιε δομές θα λαμβάνουν πάντα υπόψη τους την πρόσφυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και στην Διπλωματική Ακαδημία, ούτω ώστε αφού καταρτήσουν τους διπλωματές μα και να ξέρουν ε, πόσο θέλουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα να διαπνέουν την εξωτερική αυτή δράση και χρειάζεται αυτό να υπάρχει σε κάθε πολιτική θα πρέπει να υπάρχει μια σχετική υπηρεσία που να ασχολείται σε υψηλό επίπεδο με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να υπάρχει συντονισμός με τις εθνικές στρατηγικές. Τι θα κάνει η ψηλή εκπρόσωπος τι θα κάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα έχει κάποιον ε, ε, υφιστάμενό τη, θα ασχολείται όπως ο κύριος Σολάνα. Επίσης θα πρέπει και οι αντιπροσωπείες μας να ασχολούνται. Την περσμένη εβδομάδα η Υποπιτροπή για Ανθρωπίνα Δικαιώματα μετέβη στην Ουάσιγκτον και μεγάλη μας ικανοποίηση είδαμε ότι το θέμα αυτό είναι στο επίκεντρο του, του, του ενδιαφέροντος και θα πρέπει άρα να εξασφαλίσουμε ότι οι αντιπροσωπείε μα θα πρέπει να έχουν δεσμού με την κοινωνία των πολιτών για να ασχοληθούν αποτελεσματικά με το θέμα. Άρα, παραλαμβάνω, θα πρέπει η εξωτερική δράση να λαμβάνει υπόψη την δέσμευσή μα για προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε. Αμελίν. Από την Γαλλική Συνέλευση. Έχετε δύο λεπτά. Θα ήθελα με δύο λόγια κύριε Πρόεδρε να σας πω όσον αφορά τη θέση της Γαλλίας. Είναι κάτι το οποίο έγινε κατανοητό εδώ όσον αφορά τη συγκρότηση αυτής της νέας υπηρεσίας και θα ήθελα όμως επίσης να σταθώ στο πόσο σημαντικό είναι για μας η αυτονομία η δημοσιονομική αλλά επίσης να υπάρχει αυτονομία και όσον αφορά το προσωπικό αυτής της νέας υπηρεσίας. Επίση να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ Κομισιών και Κοινοβουλίου σε σχέση με την υπηρεσία, Δηλαδή για μα αυτό είναι αποφασιστική σημασία. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο, για να είναι πάρα πολύ σωστή η οργάνωση αυτή τη νέα υπηρεσία και θα πρέπει να δεχθούμε ότι θα είναι ιδιότυπο όργανο. Σου γένερης σύμφωνο 100% με αυτό το οποίο ελέγχθησαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά μπορώ λοιπόν να σας πω, είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για τη Γαλλία. Το ζήτημα του τι θα γίνει όσον αφορά τη διαχείριση των κρίσεων, αλλά και του διαστήματος μετά την κρίση, όπως είπε ο συνάδελφος, από την γαλλική γερουσία. Γιατί γνωρίζουμε ε, τη σημασία της Ένωσης για αυτά, για το προσωπικό. Τώρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά ε, την ε, ποσοτική πτυχή. Θέλουμε να υπάρχει ισορροπία σε σχέση με το ποιοι θα προέρχονται από τα κρατημέλη, ποιοι από το Συμβούλιο, ποιοι από την Κομισιόν. Τέλος, Πρόεδρε, θα πρέπει η υπηρεσία αυτή να έχει αξιοπιστία και για να έχει θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το χρονοδιάγραμμα. Καθυστερήσαμε, ίσως καθυστερήσαμε και πολύ σε αυτή την πρώτη φάση προβληματισμού. Σήμερα Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, πολλά προβλήματα που εκκρεμούν και περιμένουν λύση και εάν κάτι δεν κάνουμε το φθινόπωρο έχει ε, περάσει ένας ε, χρόνος μετά από τότε που ε, εξαγγέλθηκαν οι ευθυντές γραμμές και θα χάσουμε αξιοπιστία όχι μόνο και ο ένας προς τον άλλο αλλά και όλοι μαζί θα χάσουμε αξιοπιστία και προς τον υπόλοιπο κόσμο γιατί όλοι αυτό προσδοκούν να δουν τι θα κάνουμε, μας παρακολουθούν. Και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφανθεί στο δεσμευτικά, επίσης θα πρέπει να αποφανθεί ε, και συμβουλευτικά και στα πλαίσια της συναπόφασης. Όμως θα πρέπει να υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα γίνει η ψήφιση των σχετικών ε, αποφάσεων του Κοινοβουλίου. Από τη λουθόνια τώρα ο κύριος για δύο λεπτά. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, λίγες σύντομες παρατηρήσεις. Αύριο το κοινοβούλιο μας οργανώνει μία ακρόαση για το διπλωματικό σώμα και για το προσωπικό το οποίο θα ενταχθεί στο μέλλον στις υπηρεσίες της κυρίας Άστον. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι υποστηρίζουμε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σαρτσβόλσκι σχετικά με την γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα αν θέλετε. Θέλουμε μια πραγματική εξωτερική Ευρωπαϊκή Ένωση Βλέπω εδώ κάποια παραδείγματα. Έχουμε 14 ε, υπαλλήλου ε, στην Ικαράγουα και 14 υπαλλήλου επίσης έχουμε και στο Κίεβο. Έχουμε αμφιβολίες λοιπόν για το πόσο εξισορροπημένη είναι η πολιτική αυτή του προσωπικού στα, στις υπηρεσίες, στις συγκεκριμένε. Γιατί όπως και να το κάνουμε η πολιτική γειτονία ε, έχει μια κάποια προτεραιότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσπαθήσει να καταστεί το ταχύτερο δυνατόν ανεξάρτητη από τα μονοπόλια από τα οποία προμηθεύεται τις πρώτες ύλες. Ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική τα τελευταία χρόνια και υπάρχει εδώ ένα θέμα εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από το θέμα της ε, αξιόπιστης διαδικασίας προμήθειας πρώτων υλών έτσι ώστε να μην δημιουργούνται ελλείψεις που δημιουργούν προβλήματα στην αγορά. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στην πολιτική την οποία ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προς το ανατολικό κομμάτι της ε, Ευρώπης και προς το νότιο κομμάτι της Ευρώπης. Θυμίζω ότι η Μολδαβία, η Ουκρανία, η Γεωργία, οι χώρες του Νοτιού Καυκάσου θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη προσοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως είπα, Αύριο θα συζητήσουμε τα θέματα αυτά γύρω από τη δημιουργία της νέας υπηρεσίας της κυρίας Άστον. Λόζινγκ. Ευχαριστώ. Όσον αφορά την επέκταση, την περιγραφή των αρμοδιοτήτων της εξωτερικής υπηρεσίας, η ομάδα μου, η Γκουε, είναι εδώ πέρα στη μειοψηφία. Ήδη και οι συνάδελφοι από τη Γερμανική Βουλή άρχισαν κριτική στο ότι ενσωματώνονται αρμοδιότητες αναπτυξιακής βοήθειας στην υπηρεσία αυτή, αλλά δεν είμαστε στην μειοψηφία όσον αφορά την ενσωμάτωση και άλλων τομέων και βεβαίω κριτική που ασκείται και από μη κυβερνητικέ οργανώσει ή επίση στον τομέα τη αναπτυξιακή βοήθεια. Ήμουν πρόσφατα σε μια διάσκεψη και θα πρέπει να δούμε πώ θα εφαρμοστούν όλα αυτά. Αυτά θα ήθελα εγώ να προτείνω και είμαι στην ε, διάθεσή σας αν θέλετε να δούμε ποιους θα πρέπει να καλέσουμε για να μας συμβουλεύσουν για αυτά τα θέματα. Επίσης δεν ξέρω αν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το πόσο θα είναι το προσωπικό αυτές της υπηρεσίας γιατί κυκλοφορούν διάφοροι αριθμοί μεταξύ 2.000 και 6.000, 8.000 ατών και θα ήθελα να γνωρίζω εάν έχει ξεκαθαριστεί πόσο θα είναι το κόστος. Επίσης θα ήθελα να θέσω το ερώτημα από ποιους κλάδους θα προέρχεται αυτό το επιπλέον προσωπικό ε, καθώς ακούγεται πως προγραμματίζεται να είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός εκπροσώπων ε, ούτως ή άλλως ε, των επιχειρήσεων και των αμυντικών επιχειρήσεων. Θα ήθελα να γνωρίζω σε ποιο βαθμό θα υπάρχει ένα στρατιωτικό επιτελείο και είναι και θέμα αρχής εάν θα πρέπει να είναι ε, στρατιωτικοί μέλη αυτής της εξωτερικής υπηρεσίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κοπά για δύο λεπτά. Πρόεδρε. Είναι γνωστό σε όλους μας το μέγεθος του εγχειρήματος για την δημιουργία της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Παρ' όλα αυτά, είμαστε σήμερα στην τρίτη σε σειρά συζήτηση στην Επιτροπή αυτή για το θέμα αυτό και τα ίδια ερωτήματα που είχαμε στις προηγούμενες φορές παραμένουν για το θέμα του προσωπικού, το ζήτημα της γεωγραφικής εκπροσώπησης, της αναλογικής γεωγραφικής εκπροσώπησης, έτσι ώστε όλα τα κράτη-μέλη να έχουν την αντανάκλαση της δικής τους οπτικής μέσα στην υπηρεσία αυτή, δεν έχει απαντηθεί με σαφήνεια. Τα κείμενα που έχουμε δει μιλούν για κατάλληλη εκπροσώπηση των κρατών μελών. Αυτό δεν λέει στην ουσία τίποτα. Εμείς θέλουμε να δούμε πώς ε, η Βαρόνι Άστον έχει σκοπό να απαντήσει στο ζήτημα της εκπροσώψης Βορρά-Νότου, Δυτικής Ανατολικής Ευρώπης και μικρών και μεγάλων κρατών. Είμαστε σε ένα σημείο πια στη διαδικασία που χρειαζόμαστε συγκεκριμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Γιατί τότε μόνο μπορεί να καλυφθεί το αίτημα για διαφάνεια, το οποίο είναι το πάγιο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης θέλω και εγώ να προσθέσω τη φωνή μου για την ανάγκη ύπαρξης ισορροπίας στο επίπεδο εκπροσώπησης των φύλων σε αυτή τη νέα υπηρεσία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα κλείσει τη συζήτηση ο εκπρόσωπος της Βουλής της Φιλανδίας. Δύο λεπτά. Κυρία Η Φιλανδία έχει δύο α, ε, γλώσσες επίσημες και θα ε, ομιλήσω τη σουηδική γλώσσα, τη μειονοτική αν θέλετε αναγνωρισμένη γλώσσα, ε, μιας και προέρχομαι από τα νήσους Έλλαντ. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η δημιουργία αυτής της νέας υπηρεσίας. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά τεχνικά σημεία και τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες θα μας απασχολήσουν στο μέλλον αρκετά. Το θέμα είναι ότι το προσωπικό θα πρέπει να προέλθει από διαφορετικές περιοχές και είναι κάτι το οποίο θα λειτουργήσει εμπλουτιστικά θα έλεγα για την συγκεκριμένη υπηρεσία, κάτι το οποίο έχουμε ανάγκη. Ακριβώς αυτή η αντιπροσωπευτικότητα η γεωγραφική θα μας επιτρέψει να διαμορφώσουμε και μία θα έλεγα ταυτότητα ευρωπαϊκή η οποία θα καταστήσει τη δράση μας πιο αποτελεσματική και θα μπορέσουμε να αποφύγουμε έτσι τις αιμονές σε εθνικές αντιλήψεις που πολλές φορές οδηγούν σε εθνικισμούς. Σημείωσα με ενδιαφέρον αυτά τα οποία είπε και η κυρία Χάουταλα ε, σχετικά με τη σημασία τη μεγάλη που έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι σαφές ότι σε επίπεδο και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε επίπεδο Εθνικών Κοινοβουλίων θα πρέπει να καταλήξουμε σε ενιαίες απόψεις γύρω από το βάρος το οποίο θα έχουν ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εφόσον θέλουμε ε, να διαχειριστούμε σωστά τις κρίσεις οι οποίες θα εμφανιστούν στον κόσμο στο μέλλον, θα πρέπει να έχουμε συμφωνήσει εκ των προτέρων σε κάποια συγκεκριμένα θέματα πολιτικής. Θα πρέπει να μπορέσουμε να βοηθήσουμε φυσικά και τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά για να το κάνουμε αυτό, εφόσον θέλουμε να φτάσουμε σε επίπεδα εμπειρογνωμοσύνης τα οποία θα είναι χρήσιμα για την υπέρβαση κρίσεων, απαιτούνται να γίνουν πολλά. Και ίσως κάποιες εθνικές αρμοδιότητες θα πρέπει να αναλυθούν από την Ευρωπαϊκή αυτή υπηρεσία. Ευχαριστώ κυρία Νάουκλα. Κύριε Σούκα θα πάρει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για κάποια θέματα θα σας παραμένω στον κύριο Κριστόφσον γιατί ε, εγώ θα περιοριστώ στα του προσωπικού. Πρώτον, είναι σαφής η νομική βάση. 336 είναι το άρθρο της συνθήκης ε, βάσει της απόφασης που θα διέπει την αναθεώρηση του καταστατικού μας κειμένου. Τώρα, οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, κατά πόσον θα είναι η κατηγορία του προσωπικού, αυτό το οποίο θέλουμε είναι να μην εντάσσονται αυτοί στο εν τρίτον ε, της, ε, του κομματιού του προσωπικού που αντιστοιχεί σε κάθε χώρα. Το 50% από την Κομισιόν είπαμε. Αυτό όχι, δεν, δεν, δεν προβλέπεται. Ε, αντίθετα από ό,τι ελέγχθη. Επίσης, άλλη ερώτηση. Σε ποιο βαθμό το προσωπικό από κράτη-μέλη θα μπορεί να παραμείνει στην υπηρεσία. Προβλέπετε το εξή. Υπάρχει δυνατότητα συμβάσεων τετραετών που είναι εδώ να παραταθούν για κάποιο διάστημα, κάτι το οποίο εξαρτάται από το κράτος μέλος. Επομένως υπάρχει η σχετική δυνατότητα, αλλά το θέμα είναι πώς θα την αξιοποιήσουν τα κράτη-μέλη. Παρακάτω τα κριτήρια των διορισμό διπλωματών και λοιπόν υπαλλήλων είναι σαφές ότι σε αυτή την περίπτωση θα ασχίσουν τα γενικά κριτήρια, ότι δηλαδή ε, αξιοκρατικά σας υπενθυμίζω ότι τα γενικά κριτήρια του κανονισμού σημαίνει ότι ξεκινάμε αξιοκρατικά και επίσης θα προσλάβουμε όσο γίνεται περισσότερο και επί τη βάση της γεωγραφικής ισορροπίας. Άλλο. η εμπιστοσύνη. Πώς δηλαδή θα είμαστε σίγουροι το προσωπικό μας θα δίνει προτεραιότητα στα θέματα τα δικά μας και όχι στις διπλωματικές του υπηρεσίες του κράτους μέλους από το οποίο προέρχεται. Είπαμε ότι θα έχουμε αυτήν την τετραετία που επιδέχεται παράταση και γι' αυτό και θέλουμε να νιώσουμε συμβάσεις. Κάτι το οποίο είπε η ε, εκπρόσωπος της ε, Bundestag. αν δηλαδή δικαιούνται οι υπάλληλοι κοινοτικοί να επιστρέψουν στην χώρα προέλευσης. Αυτό δεν είναι πρόβλημα για μας. Αφού μιλούμε για διπλωμάτες από τα κρατη θα προβλέπετε ότι υποχρεούνται τα κρατη να διατηρήσουν τη θέση του διπλωμάτη που αποσπάστηκε στην εξωτερική υπηρεσία. Στην οποία θέση και μπορεί να επιστρέψει επίση, είχαν και άλλε ερωτήσει για θέματα τα οποία ε, θα σας εξηγήσει ο κ. Κριστόφασεν, στον οποίο θα δώσω το λόγο στη συνέχεια. Όσον αφορά την δημοσιονομική αυτονομία και τη διαχείριση του προσωπικού. Σας παραπέμπω σε αυτό που είπα στην αρχή. Η εξωτερική υπηρεσία θεωρείται ένα ιδιότυπο θεσμικό όργανο όσον αφορά το καταστατικό λειτουργία. Όχι θεσμικό όργανο με την έννοια τη συνθήκη, αλλά όσον αφορά το καταστατικό. Δηλαδή, θα υπάρχει αυτόνομη πολιτική για το προσωπικό και επικεφαλής θα είναι υψηλή πρόσωπος. Εδώ σταματώ, αλλά ξαναγυρίζω δύο λεπτά στο θέμα της γεωγραφικής ισορροπίας. Είναι αλήθεια ότι προς το παρόν δεν προβλέπονται πώς σωστά συγκεκριμένα. Ανατολή, Δύση, Βορρά, Ανατολή. Είναι αλήθεια ότι αυτό μπορεί να ρυθμιστεί με ποσότητα, αλλά προς το παρόν δεν προβλέπεται τίποτα. Εδώ ολοκλήρωσα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Σόκα. Πολύ σύντομα κύριε Κρίστοφεσεν. Όχι πάνω από πέντε λεπτά παρακαλώ. A number of issues which... Αντώνη. Κάποια ζητήματα που ίσως πάνε πέρα από τον κανονισμό του προσωπικού, να ρωτήσετε κάτι για τον χρόνο που αναφέρθηκε και στο πρώτο κομμάτι της συζήτησης και ίσως μπορώ να απαντήσω. Όπως υπόθηκε πολλές φορές, Υπάρχουν τέσσερα στοιχεία που χρειάζονται για να λειτουργήσει η υπηρεσία. Η βασική απόφαση, υπηρεσιακός κανονισμός, οικονομικό κανονισμό και ο προπολογισμό. Η ελπίδα μου και η προσδοκία μου είναι πω το τελευταίο κομμάτι του παζλ θα είναι ο προϋπολογισμός και όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα του προπολογισμού. Ελπίζω να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε σχέδιο προϋπολογισμού στα μέσα Ιουνίου, κάτι το οποίο σημαίνει πως ε, εάν όλοι κάνουν μία ανάλογη προσπάθεια θα μπορούμε να έχουμε ένα συμπληρωματικό προϋπολογισμό μέχρι την 1η Οκτωβρίου. Οπότε ω υπόθεση εργασία θα χρησιμοποιήσω την ημερομηνία 1η Οκτωβρίου και ελπίζω και τα υπόλοιπα να, είναι, να έχουν γίνει μέχρι τότε. Επίσης, θα ήθελα η βασική απόφαση να ληφθεί το συντομότερο δυνατόν γιατί αυτό σημαίνει πώς θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τουλάχιστον να προετοιμάζουμε τις προσλήψει. Δεν μπορούμε να κάνουμε προσλήψει για να ξεκινήσουμε δηλαδή συνεντεύξει κτλ και μόλις ε, έχουμε και τον προπολογισμό να προχωρήσουμε στις υπογραφές. Αυτά για το χρονοδιάγραμμα. Ε, προσλήψεις ε, και οι ανησυχίες των νέων κρατών μελών. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω Επιβεβαιώντας αυτά τα οποία είπε η κυρία Σούκα είναι πως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλέψει ποσοστώσεις αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο το παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά. Και αν υπάρχει κάτι το οποίο έχουμε ξεκαθαρίσει σε όλες αυτές τις συζητήσεις είναι πως αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί. Και γνωρίζει πάρα πολύ καλά όπως και όλοι οι άλλοι πως εάν δεν λύσουμε αυτό το ζήτημα θα έχουμε πρόβλημα. Γι' αυτό και η βασική απόφαση συμπεριλαμβάνει ένα μηχανισμό για να διασφαλίσουμε ότι αυτό το ζήτημα θα ε, το ελέγχουμε συνεχώς. Τώρα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κυρία Χάουτελα. Νομίζω συμφωνώ με αρκετά από αυτά τα οποία είπατε και με κάποιες από τις λεπτομέρειες. για την εκπαίδευση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, η εκπαίδευση των νέων διπλωματών. Δυστυχώς, όταν αρχίσαμε να προετοιμάζουμε τη σύσταση υπηρεσία, είδαμε πως δεν είχαμε προχωρήσει τόσο στην προετοιμασία. Οπότε, δώσαμε ένα, είπαμε πως σε ένα χρόνο θα πρέπει να έχουμε κανονίσει τα της εκπαίδευσης. Και εδώ πέρα βεβαίως θα αναμένουμε και τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η αναπτυξιακή πολιτική, κατά το οποίο έθιξαν αρκετοί ομιλητές. Μην ξεχνάμε πως παρά το ότι ο προγραμματισμός από ό,τι φαίνεται θα γίνει στην υπηρεσία, όλες οι αποφάσεις είναι αποφάσεις κομισιών τα πάντα θα καταλήξουν στην Κομισιόν. Αυτό το οποίο θα πρέπει να διασφαλίσουμε είναι να υπάρχει συνοχή μεταξύ του τι κάνουμε παραδείγματο χάρη στην οικοδόμηση ειρήνης σε διάφορα μέρη του κόσμου. Έχουμε περάσει δηλαδή το σημείο το οποίο θεωρούσαμε την αναδειξιακή πολιτική ως κάτι ανεξάρτητο από την ασφάλεια Υπάρχουν πολλές χώρες στις οποίες δεν θα υπάρχει αναπτυξιακή πολιτική χωρίς ε, πολιτική ασφάλειας και ε, αντιστρόφως. Βεβαίως. Και όλες οι προτάσεις ε, θα είναι κοινέ ε, προτάσεις από τον Επίτροπο Ανάπτυξη και την κυρία Άστον. να προσθέσω πως η πρότασή μας Επίσης θα καταργήσει τον τεχνητό διαχωρισμό που είχαμε μέχρι τώρα μεταξύ χωρών ΑΚΕ και λοιπόν το προσωπικό τώρα αν μου επιτρέπετε και τους αριθμούς η αφετηρία θα είναι μετατάξεις από την Κομισιόν και την Γραμματεία του Συμβουλίου όσον αφορά το επίπεδο των διοικητικών υπαλλήλων. Αναμένουμε πως οι μετατάξεις αυτές ε, θα συμπεριλαμβάνουν γύρω στα 800 άτομα. 600 ε, από τους οποίους θα είναι από την Κομισιόν. Βλέπετε ήδη δηλαδή πως ευθύς εξ αρχής υπάρχει μια... Ε, το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από την Κομισιόν. Θα εκδοθεί επίσης αύριο νομίζω μια έκθεση για την πρόσληψη του ενός τρίτου του προσωπικού. Βλέπετε πως εκεί αναμένουμε συνολικά το προσωπικό ε, το 2013 να είναι γύρω στα 1100 άτομα. 1150. Όλα τα νούμερα, τα μεγάλα που ακούτε δηλαδή, ε, συμπεριλαμβάνουν και το βοηθητικό προσωπικό και το τοπικό προσωπικό στις αντιπροσωπείες. Και κάτι ακόμα τώρα. Ε, είπατε για την Ικαράγουα και την Ουκρανία ότι έχουν τον ίδιο αριθμό. Ο, ο λόγος είναι απλός. Μέχρι τώρα οι εξωτερικές αντιπροσωπείες ε, είχαν ως κύριο βάρος την ανάπτυξη. Ε, αυτό πρέπει να αλλάξει. Και είναι σαφές πως πολλές αντιπροσωπείες Πράγματι, όπως και αυτοί της Ουκρανίας, χρειάζονται ενίσχυση. Και με συγχωρείτε αν μακρηγόρησα. Ευχαριστώ τον κύριο Κρίστενσεν. Τα τελικά συμπεράσματα, το τελικό σχόλιο θα το κάνει ο εισήγητης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ο κύριος Μπροκ. Παρακαλώ, όχι πάνω από πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποιες παρεξηγήσεις. Πρόκειται για μια υπηρεσία, δεν έχει δικές της ε, αρμοδιότητες εδώ πέρα και ο Χριστόφερσεν ξεκαθάρισε ορισμένα πράγματα. Το υβριδικό λοιπόν αυτό όργανο θα πρέπει να υποστηρίζει στο έργο της την ύπατη εκπρόσωπο στον συντονισμό των εξωτερικών σχέσεων που κατά βάση είναι αρμοδιότητα της Κομισιόν και στην εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας που είναι αρμοδιότητα του Συμβουλίου. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται στην Κομισιόν και από την Αντιπρόεδρο δηλαδή, της, της Κομισιόν και σε ζητήματα Αναπτυξιακή βοήθειας. Αν υπάρχει διαφωνία μεταξύ ενός επιτρόπου και της ε, ΥΠΑ τη εκπροσώπου θα λυθεί από το σώμα της επιτροπή. Και όταν μιλάμε για εξωτερική πολιτική πολιτική ασφάλειας, η απόφαση είναι του Συμβουλίου. Και έτσι είναι σαφές πως η δομή λήψης αποφάσεων ε, εξακολουθεί να παραμένει αναλύωτη, π.χ. όταν μιλάμε για τα εθνικά κοινοβούλια, όταν μιλάμε π.χ. στο γερμανικό σύνταγμα, είναι σαφές πως η τελευταία απόφαση ανήκει στην Γερμανική Βουλή. Αυτό δεν είναι καθόλου αρμοδιότητα της υπηρεσίας αυτής. Για να ξεκαθαρίσουμε τις φήμες. Κάτι άλλο. ο επιχειρησιακό τομέα θα χρηματοδοτηθεί από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, ο προϋπολογισμός ο οποίος υπόκειται στον έλεγχο του Κοινοβουλίου. Πρέπει, αυτό το αναφέρει και η συνθήκη, σας διαβεβαιώνω είναι σαφές. Οπότε υπάγεται και αυτή η υπηρεσία αυτή όσον αφορά τον διοικητικό της προϋπολογισμό στο ε, Κοινοβούλιο. σημαντικό νομίζω είναι το ότι θα γίνει και με τον κανονισμό του προσωπικού. Δεν έχουμε εμείς προβλήματα το 1 τρίτο να είναι από τα κράτη-μέλη. Όχι όμως από την αμυντική βιομηχανία. Είναι εθνικοί διπλωμάτες, οι εκπρόσωποι της αμυντικής βιομηχανίας υπήρχαν μόνο στις κομμουνιστικές χώρες στα Υπουργεία Εξωτερικών. Ε, εκεί ήταν ειδική των εξοπλισμών και στα Υπουργεία. Δεν ξέρω, η συνάδελφο από τη Γερμανική Βουλή, ε, δεν ξέρω σε ποιο κόμμα ανήκατε, ίσως έχετε μείνει σε κάποια τέτοια παλιά ε, μοντέλα ότι βρίσκονται εκπρόσωποι της αμυντικής βιομηχανίας στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει ε, να δούμε τώρα το εάν θα είναι το προσωπικό αυτό πάνω από το 1 τρίτο. Δεν το θέλουμε γιατί θα μπορούν να πούνε ότι εμείς είμαστε γενναιόδοροι και μπορούμε να στείλουμε παραπάνω προσωπικό. Επειδή τουλάχιστον το μισό των πολιτικών αυτών είναι κοινοτικέ, πρέπει τουλάχιστον το μισό του προσωπικού να είναι κοινοτικό επίση. Νομίζω πω με λίγη καλή θέληση, εν πάση περιπτώσει, θα βρεθεί ένα ε, καλό ε, συμβασμό εδώ πέρα. πάντων, δεν νομίζω να είναι τόσο τα πράγματα. Υπάρχει αρκετός ε, χώρος διαπραγματεύσεων. Να πω κάτι άλλο ακόμα. Κάτι το οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Μπλάουν το ανέφερε, δεν υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά περιγράφονται στο άρθρο 14, 63, 290 κτλ. Και αυτό ότι περιγράφει η συνθήκη εξακολουθεί να ισχύει. Ε, εξακολουθεί να έχει δικαίωμα επί του προπολογισμού και του ελέγχου του προπολογισμού και βεβαίως ε, μπορεί να ελέγχει και τις υποχρεώσεις ε, που δίνει η συνθήκη στην ύπατη εκπρόσωπο, δηλαδή πρέπει υποχρεωτικά να συμβουλεύεται το κοινοβούλιο. Το πώς θα εφαρμοστούν τώρα αυτά στην πράξη θα δούμε ότι θα υπάρξει μια δήλωση για το πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτό το κομμάτι της συνθήκης για να δούμε ποια θα είναι η συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και ύπατης εκπροσώπου. Είμαστε διατεθειμένοι εμεί να κινηθούμε όσο το δυνατόν ε, πιο γρήγορα γίνεται, αν είναι και στη διάθεσή μα η κυρία Άστον, για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για να συσταθεί η υπηρεσία. Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων θα ε, επέλθει όταν έχουν ξεκαθαρίσει όλα αυτά τα ζητήματα, στα οποία παίζει και βασικό ρόλο βεβαίω ο οργανισμό του προσωπικού. Οπότε δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις ε, επίσημες διαδικασίες εφόσον δεν έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία στην ε, διάθεσή μας. γιατί θα πρέπει να υπάρχει κοινοβουλευτικό όλογο και από το Ευρωπαϊκό και από τα Εθνικά Κοινοβούλια αυτή τη υπηρεσία για να εξυπηρετήσουμε και τα συμφέροντα των πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Μπρόκ, ευχαριστώ του ομιλητέ μα, την κυρία Σούκα, τον πρέσβη τον κύριο Κριστόφερσεν. Ευχαριστώ όλου σα που συμμετείχατε με τρόπο τόσο αποτελεσματικό στι εργασίε μα και στόχο μα είναι οι συναντήσεις αυτές ε, και ο διάλογος αυτός να συνεχιστεί για να έχουμε αυτή τη συνέργεια μεταξύ μας, οπότε θα έχουμε και άλλες συναντήσεις ερχόμενους μήνες, καθώς θα δούμε πώς θα συσταθεί αυτή η υπηρεσία. Θα ήθελα τώρα να σας προσκαλέσω όλους ε, να έρθετε εδώ πέρα σε ένα μπουφέ που υπάρχει έξω από την αίθουσα για να συνεχίσουμε